Dear Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξαναρχίσουμε. Και σας παρακαλώ όλους να ελέγξουμε ότι λειτουργούν οι ηλεκτρονικές κάρτες για να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Πρώτο θέμα. ψηφοφορία για τη συνδιάσκεψη COP20 Λίμα Περού. Έχουμε το ψήφισμά μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την ψηφοφορία. Τροπολογία 20. Α, όχι, ΔΕΒΕ 1. Για την παράγραφο 1. ΔΕΒΕ 1, τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Όχι. Με συγχωρείτε. Πέρας. Το αποτέλεσμα είναι ότι εγκρίνεται. Τροπολογία 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύει 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 32. Υπέρ. Όχι, λέει ο πρόεδρο. Τροπολογία 32. Δεκατέπτη δεν είχαμε ευθύσει την 31. Δεν την ευθύσαμε, επομένω ψηφίσουμε την 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 33. Υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 36 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Δεύε 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες έχουν έναν υπεράριθμο. Εντάξει. Πέρας. Όπως Αποσύρεται 37, πάμε στην 38. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 43 υπέρ κατά εποχές ΔΕΒΕΔΙΟ. DV2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να κάνουμε έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, έλα στο δούμε. Ας κάνουμε έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9-3. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 59. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 60. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 62. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τεροπολογία 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τεροπολογία 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πάλι οι σοσιαλιστές έχουν έναν υπεράριθμο. Εντάξει. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα, ΔΕΒΕ 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 68. Υπέρ. Κατά να εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 19 υπέρ κατά να εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 4 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 69 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 70. Θα ψηφίσουμε μόνο το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 112. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΔΒ10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΔΒ16 υπέρ κατά αποχές Θεωρώ ότι απορρίπτεται, αλλά να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη. Απορρίπτεται. Δεύτερη. έξι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα, τροπολογία 71. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές να επαληθεύσουμε, αλλά σας παρακολουθώ να σηκώνετε και τα χέρια. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Λέξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 75. Υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 76 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 78 υπέρ κατά εποχές να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Πέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 74. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 73. Υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. Δεύε 21. Υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 80. Υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 7 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 84 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ κατά εποχές. θα έλεγα ότι απορρίπτεται, αλλά ας κάνουμε έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 87. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 88. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 89 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 90 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα, για την 96 θα ψηφίσουμε μόνο το δεύτερο τμήμα. Για το δεύτερο τμήμα λοιπόν, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 97, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 101, υπέρ Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 102. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 41. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 98. Υπέρ κατά αποχές Αγκρίνεται. 105 υπέρ κατά αποχές Αγκρίνεται. 106 υπέρ κατά αποχές Αγκρίνεται. 104 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 109. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 110. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 111. Υπέρ. Κατά. Αποχές Αγκρίνεται. Τροπολογία 113. Υπέρ. Κατά. Αποχές Αγκρίνεται. 114. Υπέρ. Κατά. Αποχές αγκρίνεται. Τροπολογία 115. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 107 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 116 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 117 υπέρ. Κανείς. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 118. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 119. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 120. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Περνάμε τώρα. να την τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τοπολογία 4, υπέρ, κατά, εποχέ, εγκρίνεται. Έχουμε τον ΤΕΒ1, υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5, υπέρ, κατά αποχές κρύπτεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. DVJ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύε α. Α. Υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. DVB. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. DVC. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. DVD. Υπέρ. Κατά. απορρίπτεται. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ας το παληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη. Μάλιστα. Με ευρύ εκλουσία εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. ΔΒΕΝ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΔΒΗ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολόγια 13 υπέρ Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Εποχές. υπορρίπτεται. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύε και Υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. ΔΕΒΕΦ. Υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεβε ΔΕΒΕ-ΕΛ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. DVG. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. DVH. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. DVI. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. DVO υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΔΒΠ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΔΒΚ. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΔΒΑΡ. υπέρ κατά αποχές να γκρίνεται. Και τώρα, με ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία για το ψήφισμα. Il voto, avete votato tutti? Il voto è chiuso. per Πέρασε ψηφοφορίες. Εγκρίνεται το ψήφισμα 56 υπέρ, 2 κατά και 9 αποχές. Συγχαίρω όλους που συνυπέγραψαν το ψήφισμα. Πάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης, το σημείο 11. Έχουμε την ε, πρόταση κανονισμού για το in vitro διαγνωστικά τεχνολογικά προϊόντα. Απόφαση για την άνοιξη διοργανικών διαπραγματεύσεων. Δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι ο εισηγητή. Όχι. Μπορούμε να περάσουμε απευθεία στην ψηφορία. Να σα υπενθυμίσω ότι απαιτείται ειδική πλειοψηφία. 35 ψήφοι. Έχουμε μία ενιαία ψηφοφορία για την έναρξη των διαπραγματεύσεων την επιβεβαίωση φυσικά της διαπραγματευτικής εντολής της πρώτης ανάγνωσης και για τη διαπραγματευτική ομάδα που θα αποτελείται από τον πρόεδρο της Κομισιόν, τον συζητητή του Σκιώδης και για τον Επιτροπή, την Επιτροπή ΙΜΚΟ που θα γνωμοδοτήσει. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Ισχυρή εντολή, ο πρόεδρος. Και επομένω μπορούμε να πάμε στο επόμενο σημείο. Σημείο 12. Και στην περίπτωση αυτή Πρόκειται για μια διαπραγματευτική εντολή για τα τεχνολογικά προϊόντα και εδώ απαιτείται δική πλειοψήφια για την ψηφοφορία και θα ψηφίσουμε για την έναρξη των διαπραγματεύσεων και φυσικά θα επιβεβαιώσουμε και την εντολή για τη θέση στην οποία καταλήξαμε σε πρώτη αναγνώση και για τη διαπραγματευτική ομάδα που θα αποτελείται από τον πρόεδρο, τον εισηγητή του Σκιώδης, την εισηγητρία μάλλον του Σκιώδης και τον εισηγητή για γνωμοδότηση από την Επιτροπή ΕΜΚΟ. Συγητρία θέλει να πει κάτι. Όχι, άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Μάλιστα. Πλήρες Υιοθέτηση. Και πάμε στο σημείο 13 της ημερησίας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή ψηφίζουμε για την ε, κρίση σχετικά με τη σύμβαση για το διεθνές εμπόριο ειδών άγρια και χλωρίδα που αποκλείται εξαφάνιση, δηλαδή τη σύμβαση ΣΕΤΙΣ. Μια ενιαία ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πρέπει να σας ζητήσω το εξής. Με συγχωρείτε, υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Πρέπει να ψηφίσουμε εκ νέου. Άρχεται η ψηφοφορία, μπορείτε να ψηφίσετε. Ψήφισατε όλοι ή κάποιος ξεχάστηκε. Γιατί έχουμε 67 κάρτες, ε, αλλά έχουν τοποθετηθεί μόνο 64. Μόνο 64 έχουν ψηφίσει. Λήξη. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστούμε και διακόπτουμε μέχρι τις μισή. όταν θα ξεκινήσουμε το workshop για το αποθεματικό σταθερότητα της αγοράς. Σας ευχαριστώ και καλή συνέχεια.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

Uh, ladies and gentlemen, uh, good afternoon. Καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Αν μπορείτε να καθίσετε παρακαλώ και όσοι είστε στο πίσω μέρος της αίθουσα, για να μην χάσουμε άλλο χρόνο γιατί έχουμε πλήρη ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ για την κατανόησή σας. Καλώς ήρθατε ως εισηγητής του Κοινοβουλίου για την πρόταση της Επιτροπής για το επιθυματικό σταθερότητας της αγοράς για το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Όπως ξέρετε το σύστημα αυτό προτάθηκε τον Ιανουάριο και είναι κάτι ευρύτερο στα πλαίσια της ε, πολιτικής ενέργειας. Χέρι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπως ξέρετε, εκφράστηκε για τα θέματα αυτά. Το σύστημα εμπορίας εκπομπών, ETS, έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις, όχι μόνο εδώ μεταξύ των θεσμικών οργάνων, αλλά και στην κοινωνία των πολιτών. Καλωσορίζουμε την εργασία που έχει κάνει η Επιτροπή, που προτείνει λοιπόν μέτρα για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της υπερβολικής προσφοράς δικαιωμάτων εκπομπών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο σύστημα. Αυτό είναι ανταπόκριση και σε αιτήματα που και εμείς ως Κοινοβούλιο έχουμε υποβάλει για να αντιμετωπίσουμε τις διαρθρωτικές αδυναμίες του συστήματος και να λειτουργήσει όπως αρχικά είχε προβλεφθεί. Να σας πω επίσης ποια ήταν τα απορίσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 24 Δεκάτου το Συμβούλιο λέει σαφώς και επιβεβαιώνει ότι το ETS είναι ο κύριος ευρωπαϊκός μηχανισμός για να επιτευχθούν οι ενεργειακοί στόχοι της Ένωσης για την μείωση των αερίων θερμοκηπίου και λέει ότι πρέπει να υπάρχουν κίνητρα για την βιομηχανία και να διατηρηθούν αυτά τα κίνητρα χωρίς να αυξηθεί η γραφειοκρατία. Πριν υποβάλουμε σχέδιο έκθεσης ως Επιτροπή ΕΜΒΗ, πριν ξεκινήσουμε την πολιτική συζήτηση, είναι σημαντικό να ακούσουμε μια σειρά από εμπειρογνώμονες για να εξετάσουμε τα κύρια στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής και να ακούσουμε τις διαφορετικές απόψεις διαφόρων εμπλεκομένων. Όπως ξέρετε, η Επιτροπή ΕΜΒΗ θα συνεργαστεί με τους συναδέλφους της Ήτρε για το θέμα αυτό με στόχο η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας να γίνει τον προσεχή Φεβρουάριο. Ο συνάδελφός μου Αντώνιο Ταγιάννη που είναι ο εισηγητής της Ήτρε ε, ζητάει δυστυχώς συγγνώμη δεν μπορεί να παρευρεθεί. Υποθέτω ότι οι υπόλοιποι έχετε σημειώσει το σχέδιο της ε, εκθεσής του στην Ήτρε για το θέμα αυτό του αποθεματικού αγοράς ε, για τη σταθερότητα, MSR. Ευχαριστώ που μπορέσατε να έρθετε πολύ σύντομα, δηλαδή μετά εντός ε, πολύ περιορισμένες προθεσμίες να μας ε, παρουσιάσετε τις απόψεις σας. Καλώς ορίζω λοιπόν τους εμπειρογνώμονες με τους οποίους έχουμε κάνει πολύ έντονη ανταλλαγή απόψεων το τελευταίο διάστημα. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους και όδης Ματίας Γκρότε, και Ιαν Ντάγκαμ, που ελπίζω ότι δεν ξέχασαν ότι συμφώνησαν και εκείνοι να προεδρεύσουν τα επόμενα τμήματα αυτής της ε, εκδήλωσης. Γνωρίζετε όλοι ότι σήμερα το απόγευμα έχουμε την πρώτη συνεδρίαση του Κολεγίου των Επιτρόπων, της νέας Επιτροπής Έχουμε τον ε, Επίτροπο εδώ στο πρόγραμμά μας, μας είπε ότι θα έρθει, αλλά γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή, επειδή συνεδριάζει η Επιτροπή, θα καθυστερήσει. Θα έρθει λίγο αργότερα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα θα έρθει ο Χάουκε Χέρμαν να μιλήσει από το Eco Institute. Όμως να σας πω σύντομα πώς θα δείξει το απόγευμα. Στην επόμενη συζήτηση που θα προεδρεύσει ο Ματίας Γρότε θα δούμε τις επιπτώσεις ε, επί των τιμών όπου θα έχουμε τρεις ομιλητές Μάρκος Φέρντιναντ, Λούκα Κασίνη και Αντρέι Μάρκου που θα συμβάλλουν και εκείνοι. Και μετά θα έχουμε μια συζήτηση όπου θα προεδρεύσει ο συνάδελφος Ιαν Ντάγκαν και θα ακούσουμε αυτά που θα μας πει ο Τζέισον Άντερσον, Τζέσι Σκοτ, Πίτερ Μπότσεκ και Γιώργ ε, Φόρεστα. Αυτά αργότερα. Έχουμε λοιπόν ε, πολύ πλήρη ημερήσια διάταξη. Θέλουμε επίσης και οι συνάδελφοι να έχουν δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις, να κάνουν σχόλια στους εμπειρογνώμονές μας και να έχουν και εκείνη τη δυνατότητα να απαντήσουν. Παρακαλώ λοιπόν όλους τους συναδέλφους και όλους τους εμπειρογνώμονες να τηρούν το χρόνο τους. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στον Χάουκε Χέρμαν που είναι ε, ερευνητής υψηλού βαθμού στο Eco Institute, στο Αμβούργο. Ασχολείται κυρίως με τις εκπομπές στον τομέα παραγωγής ενέργειας και της βιομηχανίες που ε, είναι εντατικής χρήσης ενέργειας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, σας καλωσορίζω και σας και εγώ με τη σειρά μου όλες και όλους για να συζητήσουμε στο εργαστήριο εδώ την ε, Market Stability Reserve και το έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής. Ευχαριστώ και τους οργανωτές του ε, εργαστηρίου. Προ δύο εβδομάδων το Συμβούλιο Υπουργών έδωσε υποστήριξη για την απόφασή του για τη δημιουργία του αποθεματικού. Βέβαια δεν είναι και γραμμένες σε λίθους οι αποφάσεις του Συμβουλίου και θα πει τη γνώμη του και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς κοιτάξαμε ποια είναι τα πιο σημαντικά και ενδιαφέροντα σημεία. Θα σας εξηγήσω ορισμένες παραμέτρους που μπορεί να αλλάξουν στο μέλλον. Αυτό θα το κάνω στο τέλος της παρουσιάσεώς μου, αφού πρώτα σας δώσω, σας βοηθήσω να έχετε μια σύντομη ματιά για το μέλλον ε, των ε, πλεονασμάτων. Βλέπετε ένα γράφημα εδώ, ε, μια σύντομη εικονογράφηση των πλεονασμάτων μέχρι το 2020. Βλέπετε μεταξύ 14, 15 και 16 ότι αρχίζουν και μειώνονται, αλλά εξακολουθούμε και έχουμε υψηλή απόδοση των ε, ε, δικαιωμάτων εκπομπής, άρα δεν μειώνονται ακόμα οι, ε, οι όγκοι των δικαιωμάτων. Έχω δύο σενάρια. Ένα σταθερό και ένα με μείωση 1% και αν κάνετε το λογαριασμό μεταξύ των εκπομπών και της προσφοράς των δικαιωμάτων φτάνεται στο πλεόνασμα. Αυτό είναι το πλεόνασμα που είχαμε περίπου 2 εκατομμύρια τόνους δηλαδή το τέλος του 2013. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι ότι θα συνεχίσει το πλεόνασμα να μειώνεται στο μέλλον λόγω του λεγόμενου backloading, ε, του σοβαρού προγραμματισμού και σε ορισμένα σενάρια έχετε υψηλότερο ή χαμηλότερο πλεόνασμα, αλλά προς το τέλος της περίοδου θα αυξηθεί και πάλι το πλεόνασμα δεν γνωρίζουμε ακριβώς σε ποιο ποσό. Προδιετία όταν είχαμε αρχίσει να συζητούμε, εγώ είχα πει 1,4 δισεκατομμύρια το 2020, αλλά αποδεικνύεται ότι δεν είχα δίκιο. Η λειτουργία του αποθεματικού έχει ως εξή. Γνωρίζετε ότι θα αρχίσει το 2021, θα υπάρχει ένα ανώτατο και ένα κατώτατο ε, κατόφλιο με ένα ε, διάδρομο ε, περίφραξης, ας το πω έτσι, ένα hedging corridor, το άνω κατόφλιο 12% θα αφαιρείται και όταν τα δικαιώματα είναι χαμηλότερα, τότε θα αφαιρούνται κάθε χρόνο 100 εκατομμύρια τόνων εκπομπών. Τα ενδεχόμενα να ληφθούν μέτρα Υπάρχουν διάφορες επιλογές. Τώρα μπορεί να αρχίσει και νωρίτερα, μπορεί να αρχίσει και αργότερα η εφαρμογή. Το 2017 έχει συζητηθεί ως ε, χρονολογία αφετηρίας, όπου θα αρχίσει με ίσως 2 εκατομμύρια τόνους ε, δικαιωμάτων και να μπουν οι backloaded allowances πάλι στο σύστημα και όταν θα αρχίσει το αποθεματικό στα 900 περίπου εκατομμύρια τόνους. Και η τελευταία διαφάνεια είναι αυτή που σας δείχνω τώρα. Αυτό που μπορεί να κάνει κανείς ακόμη είναι να μειώσει αυτόν τον διάδρομο, τον περιφραγμένο διάδρομο, hedging corridor, και θα μειωθεί βέβαια και η ζήτηση για hedging στο μέλλον. Να, λοιπόν, εγώ τα είπα κιόλα. Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες και νομίζω τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο πάνελ όπου μπορούμε να συζητήσουμε τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχουν αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χέρμαν, ευχαριστούμε πολύ και που σεβαστήκατε το χρόνο γιατί έχουμε κάπως καθυστερήσει. Έτσι λοιπόν ε, θα σας ε, καλούσα να κρατήσετε με τους υπόλοιπους ε, πάνελιστ και θα καλέσω τον κύριο Ματίας Γκρότε να έρθει εδώ να προεδρεύσει για το επόμενο μέρος. von Και εγώ από πλευρά μου καλημέρα, καλησπέρα μάλλον, ευχαριστώ που ήρθατε σε αυτήν την εκδήλωση για το MSR. Το θέμα εμπορία εκπομπών το παρακολουθούμε εδώ και καιρό. Τελευταία μιλήσαμε πολύ για τον όπιστο βαρύ προγραμματισμό. Πάντα ρωτούσαμε τον αρμόδιο επίτροπο πότε θα περάσει από το κοινοβούλιο αυτό το θέμα. Μας ε, είπε τα Χριστούγεννα, αλλά δεν μας είπε ποια χρονιά. Λοιπόν, έχει κρατήσει πάρα πολύ αυτή η ιστορία. Πρέπει να εισαχθεί αυτός ο πιστοβαρής προγραμματισμός, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε κερδίσει απλώς χρόνο. Και τώρα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την ουσία της ε, κλιματικής πολιτικής, δηλαδή το εμπόριο εκπομπών. Δηλαδή όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να έχουν ε, σαφές πλαίσιο για να υπάρχει ασφάλεια επενδύσεων, για να έχουμε αυτό το ισχυρό μέσο, το βαρύ σπαθί, να το ακονίσουμε μάλιστα και να προσέξουμε να μην υπάρχουν 28 διαφορετικά συστήματα φορολόγησης. Γιατί θα μπορούσε και αυτό να προκύψει. Νομίζω ότι οι Υπουργοί Οικονομίας ε, των χωρών μας είναι πολύ δημιουργικοί. Λοιπόν, να δώσω το λόγο τώρα στους ε, ομιλητές μας. Πρώτος λοιπόν είναι ο κύριος Μάρκους Φέντλαντ. Όχι, μάλλον θα μιλήσει πρώτος ο Τόμας Ρόιτερς που θα μιλήσει για τις επιπτώσεις στις τιμές. Ευχαριστώ. Λέγομαι Μάρκος Φέρτιναν ε, και είμαι επικεφαλής ε, της ε, ανάλυσης για το ETS στο Thomson Reuters και έχουμε αναπτύξει ένα εργαλείο για να προσωμιώσουμε τον αντίκτυπο του υπομαθηματικού στη στη μέση και στην αγορά του Ανθρακά. Έχω αλλάξει πολλαπλές παραμέτρους της πρότασης και ε, βλέπετε εδώ ότι έχει αλλάξει η ημερομηνία έναρξης, ε, τα κατόφλια, τα επίπεδα των κατοφλιών. Έτσι λοιπόν αυτό θα το κάνω κατά τη διάρκεια της παρουσίασής μου και θα σας δείξω ορισμένα σενάρια. Όλα τα σενάρια που βλέπετε βασίζονται ε, στους στόχους για την ενέργεια και το κλίμα που συζητήθηκαν στο Συμβούλιο για το 2030 και δυστυχώ επειδή δεν έχουμε χρόνο, δεν θα μπω σε λεπτομέρειε, αλλά ευχαρίστω αν επιθυμείτε να το συζητήσουμε αργότερα. Τώρα, να ευχαριστήσω την προσοχή σας στην πρόταση της Κομισιόν. Καταρχήν, βλέπετε στα αριστερά ε, ε, ανάπτυξη της ε, υπερπροσφοράς, ενώ δεξιά βλέπετε τα αποτελέσματα των τιμών των ε, επιδομάτων ε, ε, δικαιωμάτων εκπομπών ε, αν έχουμε μείωση θα έχουμε μόνο μικρή μείωση στην υπερπροσφορά τώρα, όμως η επανεισαγωγή των δικαιωμάτων ε, όπως προγραμματισμού θα οδηγήσει ε, στο ε, ε, στο πλεόνασμα να αυξηθεί στο 2,3 δισεκατομμύρια το 2020, ενώ στο άλλο γράφημα βλέπουμε σιγά σιγά γύρω στο 2030 να σταθεροποιείται ε, το πλεόνασμα. Εδώ αυτό που βλέπετε με τις με τη σκιά είναι η ανάπτυξη του αποθεματικού σταθερότητας της αγοράς. Περιμένουμε το αποθεματικό να αφαιρέσει 1,3 δισεκατομμύρια δικαιώματα και κατόπιν η πρώτη, μέχρι το 2030 και κατόπιν θα αρχίσουν να απελευθερώνονται αυτά τα δικαιώματα. Βλέπετε ότι οι τιμές ε, θα κινηθούν γύρω στα 10 ευρώ για το στάδιο 3 και προβλέπεται γύρω στο 2020 μια αστάθεια στις ε, τιμές με το παθηματικό της ε, ε, όταν θα αρχίσει να λειτουργεί το 2021 και με το μειωμένο όριο περιμένουμε οι τιμές να φτάσουν το 2030 τα 35 ευρώ, να αυξηθούν δηλαδή. Βλέπετε ότι προφανώς είναι θέμα τι κάνει το αποθηματικό και θα πρέπει να δούμε και ένα σενάριο όταν δεν θα υπάρχει το MSR. Έτσι λοιπόν θα αφαιρέσουμε το πνευματικό σταθερό της αγοράς και βλέπετε εδώ μία πορτοκαλί γραμμή στο γράφημα και μας δείχνει ένα άλλο σενάριο. Έτσι λοιπόν το green είναι η πρώτη κομισιόν, το πορτοκαλί είναι το νέο σενάριο. Βλέπουμε στα αριστερά ότι αν δεν εφαρμοστεί το MSR θα δούμε ε, θα, ότι η υπερπροσφορά θα κρατήσει περισσότερο και όπως βλέπετε οι τιμές θα παραμείνουν σε πολύ χαμηλές τιμές το 2020 και κατόπιν επειδή θα ξαναμπούν αυτά τα δικαιώματα του πιστοβέρους προγραμματισμού και βλέπετε ότι επηρεάζει ε, και το μειωμένο ανώτατο όριο. Έτσι λοιπόν το MSR θα υποστήριζε την τρέχουσα τιμή που θα ήταν 9 ευρώ μεταξύ του 2020-2021 και του 2030 και θα οδηγούμαστε σε 4% περισσότερο μείωση μέχρι το 2030. Χωρίς το MSR η υπερπροσφορά θα συνεχιστεί για πολύ καιρό στο μέλλον και θα καθυστερήσει τις επενδύσεις στην τεχνολογία χαμηλού άνθρακα. Έχει γίνει μια συζήτηση να αλλάξουμε τις παραμέτρους ε, στο MSR ε, για να δούμε ποιος θα είναι ο διαφορετικός αντίκτυπος του μηχανισμού. Να σας δείξω τι θα γίνει αν ξεκινήσει το MSR το 2018, νωρίτερα δηλαδή. Αν δείτε το αριστερό γράφημα, βλέπετε αρχίζει να μειώνεται το πλεόνασμα το 2018, αλλά βλέπετε επίσης ότι η επιστροφή των δικαιωμάτων που έχουν προσταβερή προγραμματισμό θα βοηθήσει την ικανότητα του MSR να μειώσει αμέσω την υπερπρόσφορα και αν δείτε δεξιά για το γράφημα για τις τιμές, εδώ βλέπετε το ίδιο αποτέλεσμα. Έχουμε ήδη αύξηση των τιμών ήδη πριν το 2020, αλλά παραμένουν σταθερές ε, για πολλά χρόνια επειδή θα επανέρχονται τα δικαιώματα στην αγορά και θα έχουμε μόνο μερική αντιμετώπιση του προβλήματος αργότερα. Έτσι λοιπόν η επιστροφή των δικαιωμάτων ε, στην αγορά θα ε, είχε αποτέλεσμα αρνητικό στο μισαρ. Έτσι λοιπόν ε, αυτό που θα κάνω τώρα είναι να σας δείξω ένα σενάριο που έχουμε μία έγκαιρη έναρξη και τη μεταφορά των δικαιωμάτων επιστοβαρούς προγραμματισμού. Αν δείτε αριστερά βλέπετε ότι το πλεόνασμα πέφτει αμέσως όταν αρχίζει να λειτουργεί το MSR και αυτό γιατί το backloading δεν εμπλέκεται με αυτό το μηχανισμό. Και μια τέτοια πρόταση όπως βλέπετε δεξιά μας οδηγεί σε ε, μια υψηλότερη και σταδιακή εξέλιξη των τιμών. Θα σας δείξω τώρα και τον αντίκτυπο του να αλλάξουμε παραμέτρους όπως τα κατόφια ή το δικαίωμα απόσυρση. Αν παραδείγματο χάρη μειώσουμε το ποσοστό απόσυρση στο 10% από το 12% που προτείνει η Κομισιόν, μπορείτε να δείτε ότι μια τέτοια αλλαγή θα καταλήξει σε μια μικρή αλλαγή ε, στη συνολική διαδρομή και για την ανάπτυξη της οροπία τη αγορά, αλλά και για την ανάπτυξη των τιμών, για την εξέλιξη των τιμών. Μια αύξηση αυτού του ποσοστού ε, θα οδηγούσε σε παρόμοια αποτελέσματα, αλλά σε αντίθετη κατεύθυνση αν αυξήσω τα κατόφλια από αυτό που προτείνεται τώρα από τα 400 και το 833 σε 600 και σε ένα γιγατόνο, μπορείτε να δείτε ότι το μοντέλο μας ε, έχει κάποιες αλλαγές, προβλέπεται παρόμοια αποτελέσματα προς την αντίθετη κατεύθυνση προς το 2030 και σε αυτό το σενάριο ε, το αποτέλεσμα θα προέρθει κυρίως από το κατώτερο κατόφλι γιατί έχει να κάνει με το πόσο σύντομα επαναφέρουμε τα δικαιώματα στην αγορά. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι οι εναλλακτικοί συνδυασμοί του MSR μπορεί να επηρεάσουν πολύ σημαντικά το πόσο γρήγορα θα μειωθεί η υπερπροσφορά στην αγορά, ε, πώς, ποια εξέλιξη θα ακολουθήσουν οι τιμές και πόση μείωση ε, θα γίνει μέσω του ETS. Ε, βλέπουμε ότι αν αλλάξουμε τα κατόφυλλα ή το ποσοστό απόσυρσης έχουν ίσονο σημασία σε αντίκτυπο και στις ε, τιμές και στην υπερπροσφορά. Και βλέπουμε δύο χαρακτηριστικά του σχεδιασμού που είναι τα πιο, τα πιο σημαντικά για να έχουν αντίκτυπο ε, στην ισορροπία της αγοράς αλλά και τις τιμές που είναι το πότε θα ξεκινήσει το MSR και το πώς θα χειριστούμε τα δικαιώματα πιστοβαρούς προγραμματισμού. Σας ευχαριστώ. Ξαναδίνω το λόγο στον Πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φέρντιναντ, ας ακολουθήσει ο επόμενος ομιλητής. Επίπτωση του MSR και η συμπεριφορά των φορέων στην αγορά του κυρίου Τασκίνη από το Ινστιτούτο Ερευνών του London School of Economics. Έχετε το λόγο κύριε Τασκίνη. Το λέγομαι Λούκα Τασκίνη, είμαι ερευνητή στο London School of Economics και δουλεύω για το Ινστιτούτο Ερευνών Grantham. Τι θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω πώς εντάσσεται στην αγορά του MSR. Γιατί χρειάζεται να το εισαγάγουμε. Λοιπόν, πολύ βασική ερώτηση. Ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί το συζητάμε. Το πρόβλημα είναι ο σχεδιασμός της πολιτικής μας σε συνθήκες αβεβαιότητας. Όταν σχεδιάζουμε μια πολιτική και επιλέγουμε συγκεκριμένα ποσοστά ή ποσοστώσεις, στην ουσία δεχόμεθα και τις επιπτώσεις ως αναγκαίες. Και αυτό συμβαίνει γιατί δεν μπορούμε να προβλέψουμε τα απρόβλεπτα. Αυτό παρατηρούμε στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εκπομπών, Εμπορίες Εκπομπών, ETS. Υπήρξε ένα πολύ μεγάλης έκτασης απρόβλεπτο γεγονός που συνέβη που μείωσε κατά πολύ την ε, ζήτηση και άρα μείωσε και την τιμή. Πρέπει λοιπόν να σχεδιάσουμε ένα σύστημα που να μπορεί να προβλέψει ή να ανταποκριθεί σε τέτοιου τύπου απρόβλεπτες οικονομικές ε, ριζικές αλλαγές ή τεχνολογική πρόοδο. Πρώτα απ' όλα, ποια είναι η βέλτιστη εξέλιξη που θέλουμε. Ποιος είναι ο στόχος για να μπορέσουμε να αποτιμήσουμε πόσο λειτουργεί το MSR. Ας καταλάβουμε λοιπόν τι θα θέλαμε να επιτύχουμε. Ποιος είναι ο βέλτιστος στόχος. Ποια θα ήταν η βέλτιστη εξέλιξη αν είχαμε πλήρη πληροφόρηση. Αν είχαμε πλήρη βεβαιότητα και πληροφόρηση, μπορούμε να βρούμε, να βρούμε ποια είναι η τέλεια έκβαση. Ξέρουμε ποια θα είναι τα επιτόκια, ξέρουμε ότι αυτό σημαίνει ότι η μείωση θα αρχίσει αργότερα. Αν ε, δεν το λάβουμε αυτό υπόψη, η γραμμή είναι ευθεία. Προσπαθούμε λοιπόν αυτήν την βέλτιστη μείωση να την προγραμματίσουμε με βάση και το τι είναι η έννοια του πλεονάσματος. Είναι βεβαίως πολύ μεγάλο το πλεόνασμα. Αν μειώσουμε νωρίτερα, προβλέποντας ότι θα υπάρξει στο μέλλον έλλειψη, τότε θα πρέπει να δούμε πώς οι εκπομπές εξελίσσονται χρονικά. Πάντα θέλουμε να μείνουμε κάτω από τον άλλο το όριο. Τι παρατηρούμε λοιπόν, εδώ βλέπουμε τη μείωση ανά έτος, μέχρι το τέλος ε, της περίοδου που χρησιμοποιούμε για αυτήν την εξομοίωση. Και εδώ έχουμε τις εκπομπές. Εφόσον το ανώτατο όριο είναι καθορισμένο, είναι πώς θα κατανείμουμε τις προσπάθειες μείωσης και πώς θα κατανείμουμε τις εκπομπές. Ξέρουμε ότι οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε συνθήκες αβεβαιότητας για την οικονομία και για τις ε, μελλοντικές πολιτικές. Και λόγω αυτών των αβεβαιοτήτων οι επιχειρήσεις μειώνουν τη μείωση των εκπομπών τους και αναβάλουν μέχρι το τέλος της περίοδου αναφοράς. Αυτή δεν είναι η καλύτερη λύση. Δεν τη θέλουμε. Αυτό σημαίνει πως δεν θα έχουμε τα μέγιστα συγγνώμη, τα βέλτιστα αποτελέσματα που θα θέλαμε. Και αυτό βεβαίως μπορεί να είναι επίπτωση των απροβλέπτων. Και τα πρόβλεπτα δεν μπορούμε προφανώς να τα προβλέψουμε όταν σχεδιάζουμε την πολιτική μας. Ποιος είναι ο στόχος του συστήματος MSR. Επαναλαμβάνω. Όταν έχουμε εντελώς απρόβλεπτα γεγονότα, εντελώς απρόβλεπτους, απρόβλεπτους κραδασμούς, αυτό θα αλλάξει και την ε, αγορά τη ζήτηση για δικαιώματα. Θα σας δείξω αργότερα, αλλά τι θα κάνει το MSR, εδώ δεν το βλέπετε. Είναι να μειωθούν νωρίτερα οι εκπομπές. Αυτό είναι ο στόχος του MSR, εδώ το έχω εφαρμόσει, όπως το προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με βάση λοιπόν τα κατόφλια και τις τιμές που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το MSR θα δημιουργήσει λοιπόν μια έλλειψη και κάνοντας αυτό θα αυξήσει τη μείωση και θα μειώσει τις εκπομπές. Αυτό το παρατηρούμε σε αυτό εδώ το διάγραμμα. Η μπλε, ε, τα μπλε παραλληλόγραμμα είναι η βέλτιστη απόδοση, η κόκκινη γραμμή είναι η μη βέλτιστη λύση, όπου κάνουν περισσότερες εκπομπές στην πρώτη φάση εταιρείε και μειώνουν περισσότερο και εκπέμπουν λιγότερο αργότερα. Αυτό δεν είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα γιατί κοστίζει περισσότερο και το σύστημα είναι πιο αποδοτικό. Και η πιο σκούρα γραμμή που βλέπετε σε αυτό το διάγραμμα είναι η επίπτωση του MSR. Θα προσπαθήσει δηλαδή να μειώσει την καμπύλη της κόκκινης γραμμής. Θα προσπαθήσει να προσεγγίσει την καλύτερη λύση. Καταλήγοντας. Υπάρχουν αβεβαιότητες και ελλειπής πληροφόρηση και αυτό οδηγεί σε χειρότερες λύσεις. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε μια δυνατότητα να ανταποκριθούμε σε απρόβλεπτες εξελίξεις και στις τεχνολογικές αλλαγές. Γιατί αυτά τα δύο στοιχεία θα μειώσουν την αποτελεσματικότητα της πολιτικής μας. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ευέλικτοι. Το MSR ακριβώς μειώνει την επίπτωση των απροβλέπτων κραδασμών. Και μπορούμε να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτήν την ε, ε απόκληση από, ε, από τον επιθυμητό στόχο. Θα προσπαθήσουμε οι μειώσεις να γίνουν νωρίτερα. Αυτό που είναι πιο σημαντικό και το τόνισε και ο Μάρκου είναι ότι οι παράμετροι σχεδιασμού του MSR παίζουν ρόλο. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ποιες παραμέτρους πρέπει να εισαγάγουμε στο σύστημα αυτό για να λειτουργήσει καλά. Ιδιαίτερα θεωρούμε ότι τα κατόφλια απόσυρση και εισαγωγής πρέπει να είναι τα βέλτιστα για να μειώσουμε την απόκληση από τον επιθυμητό στόχο. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος Γρόντες, σας ευχαριστώ πολύ. Και ακολουθεί ο κύριος Ανδρέας Μάρκου, επικεφαλής του CEPS Carbon Market Forum. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την πρόσκληση. Είμαι πράγματι επικεφαλής του Carbon Market Forum και κάνουμε μελέτες, λίγο εδώ πιο κάτω είμαστε. Ο ρόλος μου είναι να συναγάγω κάποια συμπεράσματα και να σας βοηθήσω να κρυσταλώσετε κάποιες απόψεις και να δούμε και ποιες μπορεί να είναι οι λύσεις. Και αυτά θα δώσουν και τροφή για συζήτηση στο επόμενο πάνελ. Πρώτα, ο στόχος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας των Εκπομπών είναι να βρει ε, λύσεις για να φτάσουμε στο στόχο του 2050 που είναι 80 με 85% μείωση. Το δεύτερο ε, πράγμα που συνάγουμε ως συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει ένα σφάλμα στο σχεδιασμό του ETS. Είναι ένα δόμημα για να βελτιώσει την αγορά, έχει όμως έλλειψη ευκαμψίας από την πλευρά της ε, προσφοράς. Εφόσον δηλαδή μειώνεται η ζήτηση, κανονικά θα έπρεπε να μειώνεται και η προσφορά. Όμως εδώ το σύστημα έχει σχεδιαστεί χωρίς ευελιξία από την πλευρά της προσφοράς. Αυτό το έλλειμμα έχει επιπτώσει στη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα του συστήματος ε, εμπορίας εκπομπών. Βλέπουμε και τα, αυτά που μας έδειξε ο κύριο Στακίνης στη δική του ε, παρουσίαση. Υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες τώρα, όπως η, ο σχεδιασμός της αγοράς, η φύση της αγοράς που είναι νεαρά, σε σχέση με τη μακρά ιστορία άλλων αγορών αγαθών όπως του πετρελαίου και επίσης ότι τελικά το ETS είναι μια βραχυπρόθεσμη ματιά σε ένα μακροπρόθεσμο πρόβλημα με διαφορετικό τρόπο δηλαδή αυτή η βραχυπρόθεσμη ε, ματιά δεν προσφέρει τη λύση για την ε, επίτευξη των στόχων 2050 και επίσης αυτός ο μακροπρόθεσμος στόχος δεν θεωρείται νομικά δεσμευτικός χρειάζεται λοιπόν ένας μηχανισμός ο οποίος να συμφιλιώσει τη βραχυπρόθεσμη με τη μακροπρόθεσμη ε, προοπτική Έρχομαι τώρα στη λύση του MSR από τις παρουσιάσεις που είδαμε, που είναι μια λύση που προτείνεται για το μέρος των δημοπρατήσεων του EU ETS. Υπάρχει και ένα δεύτερο τμήμα που είναι η ανακατανομή που πάλι έρχεται από μια ιστορική βάση. Η παρουσίαση του Μάρκους Φέρντιναντ με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το MSR έχει στόχο να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στο σενάριο με MSR και χωρίς. Αλλά η διαφορά δεν είναι σημαντική. Δεν πρόκειται να ανατρέψει τα πράγματα δηλαδή το MSR. Γιατί αν εξετάσουμε την υπερπροσφορά στην αγορά φτάνει στην άνω ζώνη μέχρι το 2030 στα 800 εκατομμύρια τόνους αν το εισαγάγουμε δηλαδή το MSR όπως το έχουμε τώρα. Ε, καλά, θα υπάρχει μια φορά πέντε ετών αν το εφαρμόσουμε αργότερα. Αλλά αυτό θίγει την αξιοπιστία του ETS. Επίσης οι διάφορες παραλλαγές που προτείνονται του MSR, ορισμένες από τις παραμέτρους όπως ενωρίτερη ε, αφετηρία και εισαγωγή ή μη το, το βαρούς προγραμματισμού, επιφέρουν κάποιες αλλαγές κάποιες διαφορές, όχι πολύ σημαντικές. Μιλάμε πάλι για 2020 2025 αντί για το 2030. Δεν είναι δηλαδή πολύ μεγάλη η διαφορά. Πάλι είμαστε περίπου στα μέσα της δεκαετίας του 2020. Μεγάλη διαφορά θα προέλθει από το συνδυασμό ενωρής αφετηρίας και μη εισαγωγής του πιστοβαρούς προγραμματισμού. Και βλέπουμε ότι φτάνουμε τότε στην άνω ζώνη του φάσματος των 800 γύρω στο 2030 και τότε πραγματικά αυτό επιφέρει κάποια διαφορά γιατί από την πλευρά της αγοράς υπάρχει ένας πρόσθετος παράγοντας που πρέπει να εξετάσετε. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο το μοντέλο αντιδρά όταν υπάρχει σαφήνεια προγραμματισμού. Αυτό θα το δούμε λοιπόν, θα δούμε την επίπτωση στις τιμές νωρίτερα. Αυτή, αυτά αναμένω από την αγορά. Υπάρχει και ένα άλλο συμπέρασμα που θέλω να τονίσω και αρκετά σημαντικό βλέπουμε φάσματα τιμών. Ποτέ βέβαια δεν μπορεί να είναι κανείς βέβαιος τι θα δείξει το μοντέλο. Οι τιμές όμως δεν είναι και στρατοσφαιρικές, ειδικά αν λάβετε υπόψη ότι βρισκόμαστε στη λίστα, ότι βρισκόμαστε στη τιμή των 30 ευρώ τον τόνο. Αυτό με οδηγεί να κάνω ορισμένες προτάσεις και βέβαια ο πρόεδρος θα τις θέσει αυτές ε, υπόψη του επόμενου πάνελ. Μία από τις ερωτήσεις είναι ποιος είναι ο σκοπός του MSR, ποιο πρόβλημα υποτίθεται ότι θα επιλύσει. Νομίζω ότι είναι σαφές αυτό, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν και διαφορετικοί τρόποι ερμηνείας. Μπορεί το σύστημα MSR να επιλύσει το σύνολο του προβλήματος και χρειαζόμαστε ένα κουμπί reset έτσι ώστε να τα ξαναδούμε από την αρχή για να ξεφορτωθούμε και το συσσωρευμένο πλεόνασμα. Επίσης, αν έχουμε ένα πρόβλημα, το MSR αντιμετωπίζει το πραγματικό πρόβλημα. Αν είναι καλό το σύστημα, τότε γιατί να περιμένουμε. Ε, αν δεν είναι καλό, να μην το κάνουμε καθόλου. Να μην το εφαρμόσουμε καθόλου. Για μένα αυτό φαίνεται λογικό, λογικό το επιχείρημα. Μπορώ να κάνω και λάθος βέβαια, αλλά ας μου πούν τότε ποια είναι τα αντιεπιχειρήματα η εισαγωγή του μέτρου έχει επιπτώσει σε άλλα ε, μέτρα προστασία του περιβάλλοντος. Όπως ακούσαμε ορισμένα πράγματα δεν τα ακούσαμε όλα. Το MSR θα χρειαστεί ρυθμίσεις για να προσαρμοστεί στις νέες παραμέτρους της αγοράς, ενέργειας και ούτε καθεξής. Αν, κάνουμε, αν χρειαστεί να κάνουμε προσαρμογές, πώς θα τις κάνουμε. Και τέλος ο πρόεδρος είπε για το Συμβούλιο του Οκτωβρίου και τις αποφάσεις για το MSR. Δεν έχουν αλλάξει τίποτα στη συζήτηση όπως τη γνωρίζουμε ως τώρα. Και νομίζω ότι και αυτό πρέπει να τεθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας και τώρα θα δώσω το λόγο στους ε, συναδέλφους ε, να δούμε ποιοι ζητούν το λόγο από διάφορες ομάδες. Παρακαλώ αν μπορείτε να σεβαστείτε το χρόνο του ενός λεπτού για να μπορούν και οι προσκεκλημένοι να απαντήσουν τις ερωτήσεις. Ιβο Μπέλετ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Ματίας. Θα μείνω στο ένα λεπτό και θα κάνω δύο πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις. Ο κύριος Τακίνη Αναφέρθηκα στις παραμέτρους του MSR, του αποθεματικού Σταθερότητας της αγοράς. Είπατε στην παρουσίασή σας ε, ότι αν έχουμε κάποια κάποια κατόφλια ε, για την προσθήκη θα πρέπει να καθοριστούν και να είναι προσαρμόσιμα. Αυτό σημαίνει ότι τα επόμενα 15 χρόνια θα πρέπει να είναι ευέλικτα, δηλαδή να μην σταθεροποιηθούν. Θα πρέπει να έχουμε κάποια ευελιξία σε όλα αυτά. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Και η δεύτερη ερώτηση σε όλους ε, και στους τρεις προσκεκλημένους. Ένα από τα επιχειρήματα, κύριε Μάρκου, θα μπορούσε να είναι, και κάνω εδώ το δικηγόρο του διαβόλου, προκειμένου να περιμένουμε για την εφαρμογή το κόστος ε, για τον κλάδο, για τη βιομηχανία. Δηλαδή θα μπορούσε να αντιμετωπίσει η βιομηχανία κάποιες πάρα πολύ υψηλές τιμές που θα εκτοξευτούν και πώς, ε, πώς θα απαντήσουμε στις ενεργοβόρους βιομηχανίες της ανάγκες. Σας ευχαριστώ, ο κύριος Μιλστόλβαλτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ορισμένες ερωτήσεις σε σχέση με την θική της πολιτικής, ε, για να το αποκαλέσω έτσι. Καταρχήν, ε, ήμασταν αρκετά νοήτε για να δεχτούμε ε, το σύστημα εμπορίας εκπομπών γιατί είχαμε κάποιον πολύ έξυπνο από το London School of Economics ε, που ήρθε εδώ και μας είπε είναι τέλειο σε αυτός ο τρόπος για να λύσουμε το πρόβλημα και εμείς το πιστέψαμε. Κατόπιν πήγαμε στον οπισθοβαρή προγραμματισμό γιατί δεν λειτουργήσε το σύστημα και κατόπιν ε, ήρθαν και κάποιοι πάνσοφοι εδώ και μας είπαν να, γιατί να κάνουμε οπισθοβαρή προγραμματισμό θα λύσουμε το πρόβλημα και έξι μήνες αργότερα έχουμε έναν ε, κάποιο καινούργιο εδώ στο βήμα που ήρθε και μας λέει δεν λειτουργήσε ο οπισθοβαρής προγραμματισμός Επομένως έχουμε τώρα ένα νέο σύστημα παθηματικού σταθερό της αγοράς που θα λύσει το πρόβλημα για όλη μας τη ζωή. Αν ε, οποιοδήποτε χειραγωγούσε την αγορά, οποιοδήποτε τμήμα της αγοράς, έτσι όπως το κάνουμε εμείς τώρα. Παραδείγματος χάρη ε, την αγορά συναλλάγματος θα είχε μπει στη φυλακή. Και αυτοί τώρα οι έξυπνοι άνθρωποι από τα διάφορους ε, θεσμούς ε, θα θεωρούνταν συνεργή σε έγκλημα. Μπορείτε λοιπόν τώρα εμάς να μας βρείτε ένα κατάλληλο πολιτικό τρόπο για να βγούμε από αυτό το μπέρδεμα που έχουμε δημιουργήσει. Ευχαριστώ, Πίτερ Λίζα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές και όλους τους παρευρισκόμενους. Αυτό αποδεικνύει ότι το Κοινοβούλιο παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέταση του θέματος αυτού. Υπήρξε μία ερμηνεία από το Συμβούλιο ότι όλοι έχουν αποφασιστεί. Αλλά αυτό δεν ισχύει. Το Συμβούλιο είπε ότι πρέπει να υποστηριχθεί το σύστημα αυτό, αλλά οι λεπτομέρειες, για παράδειγμα η χρονική στιγμή εισαγωγής που συζητάμε, είναι σημαντική και είναι καλό που όλοι όσοι ενδιαφέρονται είναι αυτό. Κύριε Τόρβαλτς, για αυτό που είπατε, νομίζω ότι δεν είναι σωστή η παρουσίαση της κατάστασης. Εδώ στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή μας ήδη πολλοί το 2002-2003 είπαν ότι όπως μας προτείνεται το σύστημα αυτό εμπορίες εκπομπών από την Κομισιόν και το Συμβούλιο δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει. Κάναμε κάποιους συμβασμούς για πολιτικούς λόγους αλλά πρέπει κανείς να μαθαίνει από τα λάθη του και πιστεύω ότι δεν ήταν φυσικά όλα προβλέψιμα από τότε. Είχαν ε, προταθεί κάποιες προδιαγραφές και διαδικασίες για την ε, δημόσια πώληση, για την ε, δημοπρασία. Και το θέμα είναι μέχρι ποιο σημείο μπορούν να ανέβουν οι τιμές. Υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί. Ποια είναι μια ρεαλιστική τιμή εάν εισαχθεί η πρόταση της Κομισιόν. Ορισμένοι μιλάνε για 100 ευρώ. Αυτό βέβαια δεν είναι ρεαλιστικό. Για ποια τιμή πρέπει να... Ε, σε προς ποια τιμή πρέπει να ε, προσανατολιζόμεθα. Ποια θα ήταν μια ρεαλιστική τιμή. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος, κύριε Λίζε. Και εγώ έχω εγγραφή για να κάνω ερωτήσεις ως και συγητής. Ωραία. Άχερ τελευταίος τότε, η ερώτηση αφορά τις ε, αγορές και το ότι παρεμβαίνουμε στις αγορές. Κοιτάξτε, στις ε, χρηματοπιστωτικές αγορές, εάν αφήσουμε τα πάντα ε, στην ελεύθερη αγορά, τότε θα έχουμε πολλά προβλήματα και στο γεωργικό τομέα Επίσης παρεμβαίνουμε. Σε όλες τις αγορές παρεμβαίνουμε. Και η, αγορά, και η συζήτηση για τον οπισθοβαρή προγραμματισμό επίσης είναι σκόπιμη. Κανείς δεν λέει ότι θα είναι η λύση του προβλήματος, αλλά θα μας δώσει τον επαρκή χρόνο για να συζητήσουμε πώς θα εισαχθεί το MSR. Α, το, αυτό που με ενδιαφέρει έχει να κάνει με τη διαρροή άνθρακα. Ξέρουμε την τιμή τώρα, αλλά αυτή η διαρροή εισάγει αβεβαιότητα και θα ήθελα να μάθω πώς την αντιμετωπίζετε. Και θα ήθελα να μάθω πώς θα συμπεριλάβουμε στον υπολογισμό μας αυτή τη διαρροή άνθρακος, carbon leakage. Πώς λοιπόν θα μπορέσουμε να έχουμε πιο ρεαλιστική εκτίμηση. Ο Μπάς Άχερ τελευταίος. Ευχαριστώ Ματίας και για τα σχόλιά σου. Αν Έιλες ε, είπε πάνω κάτω αυτά που ήθελα και να πω, δεν άκουσα ποτέ να λέει ότι ο πίστοβερης προγραμματισμός ήταν μια λύση, ήταν μάλλον ε, πολιτικός συμβιβασμός, ε, για να το πω έτσι. Όμως αυτός ο πολιτικός συμβιβασμός μας δημιουργεί ένα πρόβλημα και αυτή είναι η ερώτησή μου, γιατί αν τώρα έχουμε μια λύση MSR, αποθεματικού, ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον να είναι όσο δυνατόν πιο ευφυής, γιατί για να έχει μία προβλεπόμενη εξέλιξη ε, η τιμή. Και η ερώτηση στον κύριο Φέρντιναν είναι, αν δούμε τώρα την πρόταση της Κομισιόν, καταρχήν έχουμε πιστοβερή προγραμματισμό, έτσι λοιπόν, έχουμε ε, πλεονάσμα και μετά έχουμε περισσότερο πλεονάσμα και μετά το 2021 αρχίζει να λειτουργεί το αποθεματικό. Από ό,τι καταλαβαίνετε είναι γελίο αυτό στην ανάλυση σας. Ε, ε μας δείξετε ότι αν έχουμε μία έγκαιρη υιοθέτηση του MSR, τότε θα έχουμε μία των τιμών. Ε, μπορείτε να μας πείτε κάτι περισσότερο για την ε, εξέλιξη της σταθερότητας των τιμών, αν κάνουμε αυτές τις προσαρμογές στην πρόταση της Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Φέρτιναντ. Για να απαντήσει. Δύο λεπτά. Δύσκολο θα είναι. Καταρχήν ε, για την ερώτηση του κ. Μπέλετ σε ό,τι αφορά το κόστος της μείωσης για τη βιομηχανία. Όπως ε, είδατε μέσω των μοντέλων που παρουσίασα, υπάρχει μία συνιστόσα ε, που καθορίζεται στις τιμές, ε, θα δείτε ότι θα αυξάνονται οι τιμές αν είναι πιο σφιχτή η αγορά, αλλά βέβαια με χαμηλότερες τιμές έχουμε ε, και χαμηλότερη μείωση, ενώ με μεγαλύτερες τιμές έχουμε μεγαλύτερη μείωση και υπάρχει τώρα ουσιαστικά μια διαφοροποίηση, ένα χάσμα μεταξύ της μακροπρόθεσμης εικόνας της αγοράς και της βραχυπρόθεσμης. Ε, αν λειτουργήσουμε βραχυπρόθεσμα θα δούμε, δεν θα δούμε τα σημάδια που χρειάζεται ο αγορά για να επενδύσει στι τιμέ που χρειάζεται για να φτάσει στη μακροπρόθεσμη Ό,τι αφορά τι τιμέ, σα έδειξα κάποια σενάρια. Φυσικά όλα αυτά εξαρτώνται από το ποια μορφή θα πάρει το αποθεματικό, το MSR και πώς θα εξελιχθούν άλλοι σημαντικοί παράγοντες, ποιες θα είναι οι οικονομικές εξελίξεις. Παραδείγματο χάρη, ποιοι θα είναι οι στόχοι μείωση των αερίων του θερμοκηπίου για το 2030, θα υπάρχει η αλλαγή μετά το Παρίσι του χρόνου. Έχουμε λοιπόν πολλά ερωτηματικά. Νομίζω ότι πολλή δουλειά πρέπει να γίνει ακόμη. Αλλά σε γενικέ γραμμέ υπάρχει πάντα ένα παζάρι μεταξύ του που μπορεί να πετύχει ε, τώρα και σε ένα μετέπειτα στάδιο. Και φυσικά αυτό εξαρτάται και από τι τιμέ. Και σε ό,τι αφορά την ερώτηση του κυρίου Λίσσα για τι τιμέ, εγώ σας, σας ανέφερα κάποια παράλληλα σενάρια για τους οικονομικούς δείκτες, έτσι η μέση τιμή μεταξύ του 2021 και του 2030 με την, ε, το βασικό σενάριο του ΑΕΠ 1,7 ε, μέχρι το 2020 και 1,9 μεταξύ του 2021 και 2030 είναι 24 ευρώ ανατόνο. Αυτή είναι η μέση τιμή και αν ε, έχουμε το σενάριο με ΕΚΠΑ 1% θα έχουμε 15 ευρώ για την ίδια χρονική περίοδο 2021-2030 και αν έχουμε 3% του ΕΠ που είναι αρκετά αισιόδοξο θα έχουμε 48 ευρώ ένα τόνο μεταξύ του 2021 και του 2030. Και τέλος ε, η ερώτηση για τη σταθερότητα της ε, σημερινής τιμής φυσικά πώς ορίζεται το σταθερό, από αυτό εξαρτάται αλλά νομίζω ότι σας έδειξα στην παρουσίασή μου ότι αν έχετε μία έγκαιρη ημερομηνία έναρξης του 2018 και μεταφέρετε τα δικαιώματα αμέσως στο παθεματικό, αντί να τα απελευθερώσετε και πάλι στην αγορά, θα δείτε ότι το πλεόνασμα στην αγορά μειώνεται σταδιακά, πολύ σταδιακά. Και αυτό οφείλεται στο ότι το ανώτατο όριο δεν ε, θολώνεται πλέον η εικόνα του από ε, την αγορά της υπερπροσφοράς. Βλέπετε λοιπόν ότι οι τιμές αντιδρούν. Έτσι, επομένως, έχουμε μία σταδιακή αύξηση των τιμών σε ένα τέτοιο σενάριο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Στακίνη. Σε δύο λεπτά αν μπορείτε. Ναι, να αρχίσω με το πρώτο τις προσαρμογές των παραμέτρων. Χρειάζεται αυτή η δυνατότητα προσαρμογής. Το MSR, το αποθεματικό δηλαδή, έρχεται ως συνέπεια του ότι δεν είχαμε βάλει από την αρχή αρκετή ευκαμψία στο σύστημα. Γι' αυτό εξηγεί και ο Αντρέη. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε προσαρμόσιμες παραμέτρους. Αλλά πρέπει κυρίως να κατανοήσουμε ποιος είναι ο στόχος του αποθεματικού και μετά να σχεδιάσουμε τις ε, προσαρμόσιμες αυτές παραμέτρους γύρω από αυτόν τον στόχο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση του συστήματος, του αποθεματικού, του MSR δηλαδή. Τώρα θα προσπαθήσω να υπεραμεινθώ των παλιών συναδέλφων μου του ε, London School of Economics αν προκάλεσαν κάποιο πρόβλημα, λυπούμε πολύ. Εγώ πάντως ήρθα εδώ για να προσπαθήσω να κατανοήσω ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή εντοπίσουμε το πραγματικό πρόβλημα και αυτό ε, σχετίζεται με αυτό που είπε ο κ. Γκρότε, δηλαδή η αγορά των ε, δικαιωμάτων εκπομπών καυσαέριων είναι τεχνητή αγορά. Επομένως είναι μοιραίο ότι θα παρεμβαίνουμε σε αυτήν και θα την σχεδιάζουμε. Και πάλι δεν λέω ότι το αποθεματικό θα λύσει το πρόβλημα, διότι το αποθεματικό το MSR ίσως μπορέσει να μειώσει αυτή την ε, όχι απόλυτα άριστη λύση, δηλαδή να είναι κάπως καλύτερες οι λύσεις που θα προσφέρει από αυτές τις οποίες φτάνουμε χωρίς αυτό. Ερωτήσεις τώρα που έγιναν για τις ε, παραλλαγές των τιμών. Νομίζω ο στόχος του αποθεματικού είναι να αφαιρέσει από νωρί κάποια δικαιώματα και να τα επανεισαγάγει αργότερα σε μια ανταπόκριση σε ενδεχόμενους κραδασμούς που θα υποστεί το σύστημα. Μπορείτε να τα επανεισαγάγετε αργότερα. Δεν σημαίνει ότι θα αυξηθούν αναγκαστικά οι τιμές των ε, τόνων εκπομπής. Και πάλι λέω ότι το ανώτατο όριο είναι καθορισμένο. Αν ζούσαμε σε έναν απόλυτα προβλεπόμενο κόσμο, η τιμή, η ανώτατη τιμή θα ήταν προκαθορισμένη. Και πάλι έρχομαι σε αυτό που είπε ο πρόεδρος Γκρότε. Νομίζω ότι χρειάζεται να κατανοήσουμε ότι πρόκειται για μια τεχνητή αγορά. Είναι μια σχεδιασμένη αγορά με ποσοστώσεις που εγκρίθηκαν για να επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο στόχος. Ο στόχος αυτό τώρα δεν επιτυγχάνεται λόγω της απρόβλεπτης ύφεση και ούτω καθεξή. Τέλος ο κύριος Μάρκο. Σύντομε απαντήσει μέσα στα δύο λεπτά που μου δίνετε. Ασφαλώς χρειάζεται κάποια ευελιξία Μιλάμε για ένα μηχανισμό που θα αρχίσει να λειτουργεί σε 5-6 χρόνια από τώρα. Θα χρειαστεί κάποιες προσαρμογές, κυρίως αφού θα είναι και μια νέα επινόηση, μια καινούργια μηχανή. Θα αλλάξει και η βιομηχανία. Θα αλλάξει και το επίπεδο εκπομπής ε, διοξιδίων του άνθρακα. Τώρα για αυτή την carbon leakage, δηλαδή για τη μετεγκατάσταση βιομηχανιών ε, σε χώρες που έχουν λιγότερο αυστηρούς όρους, δεν ξέρω ποια θα είναι η επίπτωσή σας, υπενθυμίζω όμως ότι έχουμε την carbon leakage list του 2020, έχουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που προβλέπουν για μετά το 2020 και πολλοί φορείς κάνουν και μελέτες για την προσαρμογή των επιπέδων παραγωγής. Αυτά πρέπει να συζητηθούν για να ληφθούν υπόψη. Όσον αφορά τώρα την τιμή αναφορά των 30 ευρώ, τα 30 ευρώ δεν αναφέρονται στις σημερινές τιμές, αλλά στο carbon leakage που στο κάτω της γραφής είναι διαρροή επενδύσεων. Και αυτό είναι μακροπρόθεσμο θέμα. Αν δεν έχουμε τα 30 ευρώ σε μια προοπτική 15-20 χρόνων, τότε έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα και αν δεν λύσουμε το πρόβλημα διότι τότε δεν θα έχουμε πλέον ε, θα έχουμε μηδενική τιμή ή θα έχουμε μια τιμή που όλο και θα φτάνει και θα φτάσουμε στα 30 ευρώ τον τόνο ε, εκπομπής. Για την τελευταία ερώτηση τώρα. Ποιος είναι ο σκοπός του αποθεματικού του MSR. Εμείς το κάνουμε αυτό για να μην χρειάζεται να κάνουμε τον οπισθοβαρή προγραμματισμό. Αυτό είναι σαφές διότι θέλουμε ένα προβλεπτό τρόπο, μηχανισμό για να αντιμετωπίζουμε τους κράδασμους. Αυτό που κάνει το MSR είναι ότι βάζει ένα χαρακτηριστικό σχεδιασμού που δεν είχε μπει στην αγορά, διότι κάνει λάθος ο κόσμος βέβαια στο σχεδιασμό των αγορών, καμιά φορά τι να κάνουμε, αλλά βοηθεί το EU ETS, το σύστημα εμπορίας δηλαδή εκπομπών, να λειτουργήσει σαν μια γνήσια πραγματική αγορά. Και υπενθυμίζω ότι ε, υπησέρχεται ιδίω στο τομέα των δημοπρατήσεων. Το ότι θα γίνει μετά από το ETS ε, όπως, η Καλιφόρνια ή το Κεβέκ κλπ. Όλες αυτές έχουν πρόβλεψη για ευκαμψία και από την πλευρά της προσφοράς. Με διαφορετικό τρόπο βέβαια. Αλλά έχουν προβλέψει διότι διδάχθηκαν από το ETS. Γιατί λοιπόν το EUTS να μην διδαχθεί και από άλλους. Ευχαριστώ για αυτές τις παρουσιάσεις και τις συζητήσεις και τις απαντήσεις σας. Το δεύτερο τμήμα λοιπόν τώρα και να δώσω την προεδρία στον συνάδελφό μου Ιαν Ντάνκαν. Ladies gentlemen, thank you very much. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ και για αυτό το τμήμα της συζήτησης. Έχουμε εδώ σήμερα τέσσερις ομιλητές που ελπίζω ότι θα επιτρέψουν να γίνει μια συζήτηση μεταξύ των ευρύτερα εμπλεκομένων γιατί ένα πρόβλημα που έχουμε είναι ότι πολλές φορές ε, μοιάζουμε απόμακροι. Λοιπόν, όσο περισσότερα μας πείτε, τόσο περισσότερο θα καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε ούτως ώστε το σύστημα εμπορίας εκπομπών ETS να λειτουργεί. Γιατί όλοι συμφωνούμε ότι δεν λειτουργεί σε αυτή τη φάση. Ποιοι είναι οι ομιλητές. Jason Anderson, επικεφαλής ε, της πολιτικής για ενεργειακά θέματα και για θέματα της Ένωσης ε, του Παγκόσμιου Ταμείου για την Άγρια Χλωρίδα και Πανίδα. Jesse Scott, επικεφαλής ε, του περιβάλλοντος του Euroelectric, είναι επικεφαλής του Euroelectric από το 2012, προηγουμένως και θέσεις στο Δήμος Europe για την ενέργεια και προηγουμένως ήταν σε μια άλλη εταιρεία ο κύριος Πίτερ Μπότσακ που είναι επικεφαλής ε, της ε, ε, ο μονάδας πολιτικής για θέματα περιβάλλοντος από την εταιρεία, από την Ένωση συγγνώμη, των Ευρωπαϊκών Βιομηχανικών. Ο κύριος Ντεκ Φόρεστερ είναι πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης ETS. Ο καθένας θα μιλήσει για έξι περίπου λεπτά και μετά ε, όλοι οι εκπρόσωποι εμπλεκόμενων και ενδιαφερομένων φορέων θα μπορούν να έχουν τον λόγο. Σας παρακαλώ όταν θα πάρετε τον λόγο να μας παρουσιάσετε το βιογραφικό σας σύντομα και να περιοριστείτε στο θέμα που έχουμε για να αξιοποιήσουμε τον ε, χρόνο μας. Δεν θα πω πολλά για την δική μου θέση. Αλλά πρέπει να πω ότι είναι κρίσιμη συγκυρία. Εάν διορθώσουμε τώρα τα πράγματα, δεν θα τα διορθώσουμε ποτέ. Α ακούσουμε λοιπόν του εμπειρογνώμονε. Jason Anderson λοιπόν πρώτο. Παρακαλώ. Jason. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Χαίρομαι που είμαι παρόν. Θα είμαι σύντομο, ίσω και λιγότερο από 6 λεπτά. Γιατί με βοηθάει αυτό το έγγραφο με τις θέσεις μας, εκεί πίσω υπάρχουν αντίγραφα Έχω συνεργαστεί με τους εταίρους μας, Market Watch, Greenpeace και Sandbank, όλοι μαζί υπό την αιγίδα της οργάνωσης ε, δράση για το κλίμα στην Ευρώπη, για το MSR. Να αναφέρω μερικά από τα κύρια σημεία. Γιατί η κοινότητα αυτών που ασχολούνται με το περιβάλλον ενδιαφέρεται τόσο πολύ για ένα τόσο τεχνικό θέμα. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο δημιουργήθηκε το ETS από τότε που υπήρχε το πρόγραμμα για την κλιματική αλλαγή της Ένωσης πριν από το 2003 και έχουμε παρακολουθήσει ένα σύστημα. Στην αρχή στα βρεφικά του πρώτα βήματα είχε πολλά προβλήματα παιδικών ασθενειών και όταν ε, υπήρχαν κάποια προβλήματα έτσι βρεφικά ας πούμε, κακή συμπεριφοράς βρέφους Εντάξει, ήμασταν επικείς, αλλά τώρα έχει περάσει σε εφηβική ηλικία και υπάρχει πολύ ε, ευρύ χάσμα μεταξύ αυτού που μας λένε τα όργανα της Ένωσης για το πώς θα έπρεπε να είναι υποδειγματικός έφηβος και την πραγματικότητα της συμπεριφοράς του. Μήπως λοιπόν πρέπει να πάει σε αναμορφωτήριο. Το MSR λοιπόν είναι απόλυτα αναγκαίο αλλά όχι ικανό, σίγουρα, αυτό θα το πω. Λίγο παρακάτω. Έχουμε μια σειρά από προτάσεις που μπορείτε να δείτε σε αυτό το έγγραφο των θέσεών μας. Πρώτη, και από αυτού νομίζω ότι όλοι οι παρατηρητές συμφωνούν, είναι ότι το MSR πρέπει να ξεκινήσει νωρίτερα. Εμείς προτείνουμε να ξεκινήσει το 2016. Τώρα αρχή μέσα του 2016, μέσα του 2017. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να μπορέσει να αντιδράσει καλύτερα στα στοιχεία που θα έχουμε τον Μάιο του 2016 και το 2021 να έχουμε αναθεώρηση, άρα ε, πέντε χρόνια νωρίτερα από ό,τι προβλέπετε. Τώρα, γιατί είναι σημαντικό να ξεκινήσει τώρα το πρόγραμμα. Δεν έχουμε ένα θεωρητικό πρόβλημα για το οποίο θέλουμε μια τεχνική λύση. Το πρόβλημα υπάρχει τώρα και το πρόβλημα θα οξυνθεί από κάτι άλλο που σήμερα ακούσαμε και για το οποίο είναι εντυπωσιακό ότι όλοι συμφωνούν ότι η, ε, τα δικαιώματα που βαρός θα εισαχθούν δεν πρέπει να αφαιρεθούν γιατί θα έχουμε και 800 εκατομμύρια και παραπάνω. Άρα δεν θα αντισταθμιστούν. Στην ουσία λοιπόν θα μεγαλώσει πάρα πολύ το αποθεματικό. Επίσης, ακούσαμε ότι πρέπει να γίνουν τεχνικές αλλαγές στο ανώτατο και κατώτατο όριο και να μειωθούν αυτά τα όρια στο μέλλον. Είναι λογικό λοιπόν και αυτό το διάστημα μεταξύ των ε, δύο ορίων πρέπει να ε, μειωθεί σταδιακά. Είδαμε διάφορα διαγράμματα σήμερα που μας λένε ότι θα ε, αλλάξει ε, δραστικά η τιμή του το 2030. Δεν θέλουμε λοιπόν αυτές οι εξοικονομήσεις σήμερα να μετατραπούν στο μέλλον σε μαζικές δυνατότητες μόλυνσης. Πρέπει να υπάρχει όριο λοιπόν στον αριθμό των δικαιωμάτων που μπορούν να μεταφερθούν. Αυτό το MSR πρέπει ακριβώς όπως λέει και ο τίτλος του να μας χορηγήσει σταθερότητα. Αλλιώ θα είναι δαμόκλειος σπάθη η ύπαρξη τόσων δικαιωμάτων σε ένα παθηματικό. Αυτό είναι τμήμα της λύσης για τα προβλήματα του ETS. Θα δούμε τι περαιτέρω νομοθετήματα θα γίνουν εντός του ε, πλαισίου για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υπερβολικής προσφοράς. Και το θέμα είναι ότι οι προβλέψεις για το ποσό της υπερπροσφοράς μπορεί να είναι υποτίμηση του προβλήματος. Θέλουμε λοιπόν να μειώσουμε τα προβλήματα που είχαμε στο μέλλον. Δεν είχαμε φανταστεί τι θα μπορούσε να συμβεί αν υπήρχε ε, ένα συγκεκριμένος αριθμός δικαιωμάτων στο σύστημα. Και μπορεί να μην είναι δύο, αλλά τέσσερα δις. Γιατί βλέπουμε ότι μέσω ανανεωσίμων και απομάκρυνση από τον άνθρακα ήδη μειώνουμε τις εκπομπές. Άρα θέλουμε συνολικά να υπάρξει πολύ πιο φιλόδοξη πολιτική απομάκρυνση από τον άνθρακα. Και τέλος, πρέπει να αντιμετωπίσουμε και διαρροή άνθρακα, που να είναι ρεαλιστική. Δηλαδή από τη μία ο να πληρώνει, αλλά να δημιουργηθεί ένα ουσιώδες σύστημα κινήτρων για καινοτομίες στην Ευρώπη. Δεν πρέπει λοιπόν να το βαρύνουμε μέσω του MSR. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστώ πολύ κύριε Άντερσον. Ελπίζω ότι είναι μπορέσουμε να στείλουμε στο αναμορφωτήριο το σύστημα εμπορία εκπομπών. Κατόπιν ε, κύριο Σκοτ. Κυρία Σκοτ, ευχαριστώ. Είμαι εδώ από τη Euroelectric ε, που εκπροσωπεί τον Ευρωπαϊκό τομέα ηλεκτρική ενέργειας, αλλά και ω τμήμα ενό ευρύτερου συνασπισμού επιχειρήσεων. Έχει κυκλοφορήσει αυτή η επιστολή με 59 λογότυπα και καλή για να αναλάβουμε έγκαιρη δράση για τη μεταρρύθμιση του MSR. Αυτό ο συνασπισμό καλύπτει ε, πολλούς τομείς, 4,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και νέα 3 εκατομμύρια περιουσιακό στοιχείο, γιατί έχουμε πάρα πολλά ε, και μεγάλους επενδυτές και επίσης ε, υποστηρίχθηκε από αυτό το συνασπισμό το backloading ε, του ETS. Ξέραμε όμως ότι δεν ήταν μια λύση. Εμείς θεωρούμε ότι το αποθεματικό σταθερό της αγοράς μπορεί να αποτελέσει μια λύση και το υποστηρίξαμε για παρόμοιους λόγους για αυτούς που η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλες κυβερνήσεις το υποστηρίζουν θέλουμε ε, αποθεματικό σταθερό της αγοράς ε, πριν το 2020. Εμείς θα θέλαμε να ξεκινήσει το 2017 διαφορετικά. Όπω είπαν και οι αναλυτέ θα δούμε τα δικαιώματα του επιστοβαρού προγραμματισμού να ξαναμπούν στην αγορά από το 2017-2018 και κατόπιν θα δούμε ένα αποθεματικό που θα αρχίσει να προβαίνει σε αποθεματοποίηση. Και αυτό είναι ένα zigzag. Ε, και ένα zigzag φυσικά δεν μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση τη εμπιστοσύνη αγορά σε μια ευθρεστή αγορά. Αν το κάνετε αυτό, πρέπει να ξεκινήσετε τη στιγμή που το backloading, ο επιστοβαρή προγραμματισμό θα ξαναγίνει real reloading. Υποστηρίζουμε το παθηματικό σταθερό της αγοράς να ξεκινήσει νωρίς στο πλαίσιο της υποστηρίξης το στόχο 40% της μίας των νωρίων θερμοκηπίων που υποστηρίχθηκε από το Συμβούλιο με το ETS ως το κύριο μέσο παράδοσης των στόχων. Το ETS, το σύστημα εκπαιδεύσης εκπομπών, ε, ουσιαστικά εξυπηρετεί τις τρόχους. Μπορούμε να έχουμε φορολογία του άνθρακα και θέτουν τιμές προβλέψιμες. Το πρόβλημα με τη φορολογία του άνθρακα είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε έναν νέο φόρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχουμε 28 και φαντάζομαι ότι θα είναι 28 διαφορετικοί και αυτό φυσικά έχει επιπτώσεις για όλη την αγορά ενέργειας, στην εσωτερική αγορά στην Ευρώπη. Η άλλη επιλογή είναι να εισαγάγεται κάποια πρότυπα επιδόσεων, δηλαδή ανάλογα με το χαρτοφυλάκιο κτλ. Και είναι πολύ λιγότερο ευέλικτο προ την αγορά. Έτσι, από την επιχειρηματική σκοπιά, εμεί χρησιμοποιούμε μια αγορά ανθρακά, δηλαδή έναν ευέλικτο μηχανισμό τιμών. Και επίση ε, το ETS ε, όχι μόνο δημιουργεί, στέλνει ένα μήνυμα για τη μείωση των εκπομπών, αλλά έχει καταστεί και ένα παγκόσμιο μοντέλο και ξέρω ότι ο συνάδελφο θα πει περισσότερα και επομένως έχει τη δυναμική να προωθήσει την παγκόσμια διαδικασία για τη μείωση των κομπών με τη σύνδεση με τις αγορές άνθρακα που αναπτύσσονται στην Κίνα και αλλού. Και φυσικά παράγει και έσοδα τα οποία μπορούν να επενδυθούν εκ νέου στην καινοτομία χαμηλής τεχνολογίας άνθρακα τεχνολογίας χαμηλού άνθρακα. Όμως σήμερα έχουμε τρία κυρία προβλήματα που πρέπει να λυθούν αν θέλουμε να έχουμε αξιοπιστία στην αγορά. Αυτό είναι το κύριο μέσο για να φτάσουμε στο 40% και να έχουμε και αντίκτυπο στις αποφάσεις, τις επενδυτικές του κλάδου. Καταρχήν, το πρώτο πρόβλημα είναι το πλεόνασμα που αντιμετωπίζουμε σήμερα στα δικαιώματα. Εδώ έχουμε πάρα πολλά νούμερα. Ε, το αριθμό κομισιών πάνω από 2,5 εκατομμύρια το 2020 είναι τεράστιο αριθμό Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν πρόκειται για μια πραγματική αγορά. Η προσφορά είναι σταθερή, φυσικά η ζήτηση αλλάζει στον πραγματικό κόσμο. Χρειαζόμαστε κάτι που θα επιτρέψει στην προσφορά να προσαρμοστεί στην ζήτηση που θα αλλάζει. Το τρίτο πρόβλημα είναι το σημερινό ανώτατο όριο ε, δεν συνάδει με του στόχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2030. Το MSR θα λύσει τα προβλήματα 1 και 2. Το τρίτο πρόβλημα είναι για το πακέτο 2030 και θα αντιμετωπιστεί μαζί με όλα τα θέματα που αφορούν και τη διαρροή του άνθρακου. Όμω αυτό δεν είναι τμήμα του MSR. Αντιμετωπίζει το πλεόνασμα και το πρόβλημα της ευελιξίας της προσφοράς. Τώρα, ο στόχος ε, του ETS και το τελευταίο σχολείο μου είναι να πυροδοτήσει αλλαγές στα χαρτοφυλάκια και στις διαδικασίες των εγκαταστάσεων στις βιομηχανίες που συμμετέχουν, στους κλάδους που συμμετέχουν. Αν θέλουμε να έχουμε αλλαγή θα πρέπει να κάνουμε επενδύσεις και για να κάνουμε επενδύσεις το ηχηρό μήνυμα από το δικό μου κλάδο τα τελευταία πέντε έτη ήταν ότι έχουμε μια πολύ αργή και καθυστερημένη συζήτηση για το ETS και το μήνυμα ήταν ότι χρειάζεστε να στείλετε ένα ηχηρό μήνυμα πολιτική. Το καλύτερο δυνατό μήνυμα προέρχεται από το σύστημα εκπορία εκπομπών. Όμω, η σημερινή τιμή, 6 ευρώ, δεν είναι ένα μήνυμα πολιτικής και μία τιμή που θα παραμείνει εκεί, ίσως λίγο ψηλότερη το 2021, δεν είναι μήνυμα πολιτικής. Οποιοδήποτε καθυστέρηση στη μετέπειτα με σημαίνει ότι καθυστερείται και τις επενδύσεις που χρειάζεται οποιαδήποτε άλλη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα. Για το θέμα των παραμέτρων, των τεχνικών λεπτομεριών, που συζήτησε το προηγούμενο πάνελ, Έχουμε εκεί πάρα πολλέ αναλύσει, όμω οι γενικέ γραμμέ ε, ω κλάδο πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι εγχείρημα όπου θα μάθουμε μέσα από την πράξη τι είναι μια αγορά και συμμετέχοντα στην αγορά θα απαντήσουν και θα δούμε πώ θα απαντήσουν, πώ θα ανταποκριθούν. Έτσι λοιπόν ένα άλλο στοιχείο τη θέση μα είναι μια ρήτρα αναθεώρηση για το αποθεματικό πέντε έτη μετά την έναρξή του. Σα ευχαριστώ. Ο πρόεδρος Ντάνκαν, σας ευχαριστώ. Πραγματικά τηρήσατε απόλυτα το χρόνο σας. Ακολουθεί ο Πέτερ Μπότσεκ. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε που μας προσκαλέσατε. Είναι, είμαστε σημαντικοί stakeholders βέβαια για τη συζήτηση αυτή. Μιλούμε για τους κλάδους μας, για τις ε, βιομηχανίες έντασης ενέργειας που πληρώνουν το τίμημα εμείς, ε, μάλλον, εμείς βρισκόμαστε σε παγκόσμιο ανταγωνισμό και για μας οι τιμές αυτές είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Οι Αμερικανοί βουλευτές επιμένουν τώρα η Κομισιόν να παρέμβει στην ε, αγορά γιατί σας είπαν ότι το backloading δεν μπορεί παρά να είναι εφάπαξ μέτρο και το θετικό στοιχείο είναι ότι θα εισαχθεί κάποια ευκαμψία σε αυτή την αγορά, η οποία ήταν αρκετά ακαμπτή από την αρχή. Αυτό μας φαίνεται θετικό και είναι και αυτό που ζητούν οι βιομηχανίες έντασης ενέργειας από την αρχή. Εμείς είπαμε εξοπλίστε μας με τον αριθμό δικαιωμάτων που χρειαζόμαστε, δεν θέλουμε παραπάνω από αυτές που χρειαζόμαστε, παραπάνω δικαιώματα από αυτά που χρειαζόμαστε και είπαμε μάλιστα ακόμη ότι αν δεν, χρειαστού, αν δεν τα χρειαστούμε τα δικαιώματα, μην μας τα δώσετε. Μιλώ λοιπόν τώρα για ε, ευκαμψία της προσφοράς βασισμένο σε benchmark. Βασισμένη σε benchmark. Έχετε κάποιο στοιχείο εκ των υστέρων διορθώσεως όταν κλείνετε για παράδειγμα ένα εργοστάσιο χάνετε το δικαίωμα να λαμβάνετε δικαιώματα εκπομπής. Επίσης όταν μειώσετε την παραγωγή σας κάτω από ένα κατόφλι μειώνονται τα δικαιώματα εκπομπών αυτή η ευκαμψία όμως είναι πάρα πολύ περιορισμένη και εκεί μπορεί να υπάρξει βελτίωση. Τώρα που έχουν πέσει απάνω σας όλοι αυτοί οι forecaster με όλες αυτές τις προβλέψεις δεν μπορείτε τελικά να συγκρίνετε. Ένας προηγουμένως σας παρουσίασε την υπόθεση ότι οι εκπομπές του 2013 θα παραμείνουν περίπου σταθερές. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει οικονομική ανάκαμψη. Και αυτό είναι ιδιαίτερα λυπηρό. Ο άλλο λέει α βασιστούμε στην υπόθεση ότι θα είναι λίγο παραπάνω από 1% η ανάπτυξη. Θα δυσκολευτείτε πολύ να τα συγκρίνετε και να τα κατανοήσετε όλα αυτά και να τα βάλετε σε κάποια οπτική και προοπτική. Εγώ θέλω να θέσω υπέψη σας τώρα ότι υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, πάρα πολλά ερωτηματικά που δεν απαντώνται για την ώρα. Δεν γνωρίζουμε τι ε, θα προκύψει από την COP21 του Παρισιού, τη διάσκεψη για το κλίμα. Δεν γνωρίζουμε, ακόμα δεν έχουμε δει μελέτη αντικτύπου που να βασίζεται σε μια ε, ε, ε εισαγωγή του MSR. Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι είδους επίπτωση θα έχει το αποθεματικό στις τιμές του τόνου. Ένα πράγμα είναι βέβαιο. Θα, αυξήσει, θα αυξήσει, θα σπρώξει προς τα πάνω την τιμή. Δηλαδή θα επιφέρει σπάνιδα και επομένως θα αυξήσει τις τιμές. Κάποιο στοιχείο λείπει όμως. Τι γίνεται με την διαρροή των βιομηχανιών. Α, μας είπαν, με αυτά θα έρθουν αργότερα. Ας κάνουμε πρώτα το πρώτο αυτό βήμα και μετά θα δούμε. Το Συμβούλιο είπε κάτι για το Carbon Leakage Protection μετά από το 2020. Αλλά δεν μας ικανοποιούν αυτές οι προοπτικές που μας δίνεται. Εφόσον υπάρξει παρέμβαση στην αγορά θα θέλουμε, θα θέλουμε να δούμε εκ παραλίλου ταυτόχρονα ανταπόκριση στις ανησυχίες μας για την διαρροή άνθρακος, για την ε, μετεκατάσταση βιομηχανιών που δεν πρόκειται να βελτιωθεί η κατάσταση και θα συνεχίσει ως έχει. Εμείς λέμε λοιπόν ότι θα πρέπει να βαδίζουν εκ μια αύξηση της ευκαμψίας των ε, δικαιωμάτων, της προσφοράς δηλαδή, και το ETS να είναι ισχυρό απέναντι και στην ανάπτυξη. Να μιλήσουμε για ανάπτυξη, να μιλήσουμε για απασχόληση, όχι μόνο για κράδασμους. Τα όσα ακούσαμε ως τώρα θα οδηγήσουν σε αύξηση και της τιμής της ενέργειας, όχι μόνο για τη βιομηχανία, αλλά και για τον τελικό καταναλωτή. Ήδη σε ορισμένε χώρες μέλη έχουμε σημαντικά προβλήματα ε, φτώχειας ενέργειας. Άνθρωποι δηλαδή που δεν έχουν αρκετή ενέργεια για να ζεσταθούν το χειμώνα. Εμείς λέμε λοιπόν, ναι, μπορεί να βελτιωθεί το σύστημα εμπορίας εκπομπών και μάλιστα εμείς έχουμε και καλές ιδέες και αν μας το επιτρέψετε θα το κάνουμε διαμιάς, εφάπαξ με περισσότερη ευκαμψία για την κατανομή. Μπορούμε να το κάνουμε. Εξαρτάται από εσά αν θα μας το επιτρέψετε με το αποθεματικό. Με αυτό το εργαλείο του αποθεματικού. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπόρτσεκ. Και τώρα ο τελευταίο μα ομιλητή ο πρόεδρος ε, της Διεθνούς Επιτροπής ε, Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπαμπών, ο κύριο Φόρεστα. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ευχάριστο είναι για να σας δώσω λίγο την άποψή μας. Είμαστε επαγγελματικός οργανισμός που ασχολείται με τις αγορές εκπομπών και στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στόχος μας είναι οι αγορές να αποτελέσουν τη λύση για τα προβλήματα των, της κλιματικής αλλαγής δεν έχουμε καθόλου ελαφρύ αντιμετώπιση του θέματος. Πριν από δύο χρόνια ήμουν υπέρ εδώ παρών του οπισθοβαρούς προγραμματισμού αλλά μόνο εάν υπήρχαν συνοδευτικά διαφορετικές μεταρρυθμίσεις και σε ένα πλαίσιο ενός προγράμματος όπου το ETS θα ήταν στο επίκεντρο. Θέλουμε λοιπόν να είμαστε συνεπείς στην αντιμετώπιση μας. Θεωρούμε ότι ο πιστοβαρής προγραμματισμός θα ήταν ένα αρχικό βήμα, αλλά θα έπρεπε να είναι συνοδευόμενο. Και εξετάσαμε μια σειρά από εναλλακτικέ λύσεις για το πώς να αντιμετωπίσουμε το πλεόνασμα που υπάρχει. Να μην του κάνουμε τίποτα μέχρι να το καταργήσουμε. Να καταργήσουμε ένα μεγάλο τμήμα του. Και τα μέλη μας, η οργάνωσή μας ε, έχει το ακρονίμιο ΑΕΝΤΑ, η οργάνωσή μας λοιπόν θεώρησε ότι η εισαγωγή αυτού του συστήματος είναι μια ενδιάμεση λύση. Παίρνουμε αυτό το πλεόνασμα και να τη οξιοποιήσουμε με πιο καλό τρόπο μακροπρόθεσμα. Πώς λειτουργούν οι αγορές ε, εμπορίας εκπομπών. Γιατί υπάρχει μια διαφορά στο χρονισμό. Οι επιχειρήσεις προγραμματίζουν τις επενδύσεις τους μακροπρόθεσμα, ιδιαίτερα οι μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις, οι μεγάλες επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρισμού, 15, 20, 30 χρόνια. Αλλά Πώς συμμετέχουν στην αγορά εκπομπών. Οι περισσότερες ε, περίοδοι εμπορίας είναι τριετής. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι δυνατόν ε, να αγοράσουμε τώρα γιατί δεν είναι δυνατόν. Θα ήταν πολύ ακριβό να αγοράσουμε τώρα. Και ορισμένοι έχουν προβλήματα ρευστότητας. Αλλά στα πλαίσια της δικής τους διαχείρισης κινδύνων δεν το κάνουν. Άρα υπάρχει αυτή η έλλειψη σύνδεσης. Και εσείς ως ε, κοινοβουλευτικοί που έχετε την υποχρέωση διαχείρισης ε, του δημόσιου δυναμικού ε, θα συμφωνούσατε ότι αν εισαγάγατε περισσότερα δικαιώματα σε μια αγορά όπου ήδη υπάρχει υπερπροσφορά δεν είναι καλύτερη λύση. Άρα η δομή αυτή ενός MSR για να αντιμετωπίσουμε τις ακραίες καταστάσεις αφαίρεσης από δημοπρατήσεις ε, δικαιωμάτων τώρα που υπάρχει υπερπροσφορά για να τις αξιοποιήσουμε αργότερα που θα υπάρχει έλλειψη είναι καλή λύση. Έτσι έχουμε και στρατηγικά αποθέματα αργού πετρελαίου για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενα ελλείψεων. Δεν έχουν βέβαια τιμές κατοφλίου, αλλά είναι δί να αντιμετωπίσουν προβλήματα στον εφοδιασμό. Είναι λοιπόν μια χρήσιμη παρομοίαση νομίζω για το πώς πρέπει να λειτουργήσει αυτό το αποθεματικό. Όλα έχουν να κάνουν με την χρονική αντιμετώπιση και πώς ε, στα πλαίσια του χρόνου διαχειριζόμεθα τα δικαιώματα. Τώρα, κοιτάζοντας ε, στην επόμενη δεκαετία, δεν θα μας εξέπλησε εάν αντιμετωπίσετε το αντίθετο πρόβλημα κάποια στιγμή μέσα στην επόμενη δεκαετία να υπάρχει ένα πρόβλημα δηλαδή στην προσφορά δικαιωμάτων για κάποιους απρόβλεπτους λόγους και όλοι θα θεωρούσαμε τότε ότι να πουλάμε πολύ φτηνά 6 ευρώ τον τόνο τώρα τα δικαιώματα δεν είναι πολύ καλή ιδέα. Γι' αυτό θέλουμε αυτό το αποθεματικό. Μας δίνει ένα μέσο για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα που έχουμε τώρα με ένα καλό μακροπρόθεσμα τρόπο. Συμφωνώ με ορισμένα που υπόθηκαν ήδη. Εμείς ως οργάνωση, η ΑΕΝΤΑ, μελετήσαμε τις αναλύσεις του Μάρκου και, άλλους, και άλλων και θεωρούμε ότι έχει έννοια να εφαρμοστεί νωρίτερα και ότι θα ήταν καλύτερα αυτές οι, αυτά τα δικαιώματα οπισθοβαρούς προγραμματισμού να μπουν στο αποθεματικό. Αυτή είναι μια αλλαγή που θα στηρίζαμε. Πιστεύουμε επίσης ότι βεβαίως ε, οι τεχνικές παράμετροι του συστήματος χρειάζονται περισσότερο διευκρίνηση. Και εμείς είμαστε σε φάση εξέτασής τους. Αλλά νομίζουμε ότι οι αρχικές ε, τιμές που προτείνει η Κομισιόν είναι λογικές. Τώρα να σας πω λιγάκι πώς λειτουργεί και η παγκόσμια αγορά. Το είπε και ο Άντρε Μάρκου προηγουμένως. Δεν είστε μόνοι και οι πιο πρόσφατες ε, αγορές εμπορίων έχουν χρησιμοποιήσει τέτοια αποθεματικά, όπως για παράδειγμα η Καλιφόρνια και το Κεμπέκ. Έχουν αποθεματικά για να αντιμετωπίσουν ε, ενδεχόμενα μεγάλης πτητικότητας τιμών και για να διαχειρίζονται την ροή εισαγωγή στην αγορά των δικαιωμάτων. Λειτουργούν διαφορετικά και δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν να λειτουργήσει στην Ευρώπη, γιατί έχουν κατόφλια ε, τιμών που είναι πολύ ψηλά. Μπορεί να εισαχθούν στην αγορά εάν η τιμή φτάσει τα 40, 45, 50 δολάρια τον τόνο. Άρα πρέπει να είναι πολύ ακραίες οι περιστάσεις. Νομίζω ότι η προσέγγιση της Κομισιόν που το αντιμετωπίζει περισσότερο ως θέμα προσφοράς είναι πολύ πιο κατάλληλο για το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φόριστερ και πάλι σεβαστήκατε το χρόνο. Τώρα έχουμε περίπου ένα τέταρτο διαθέσιμο για τις ερωτήσεις, όμως ο κύριος Γκρότε μόνο θέλει να κάνει μια ερώτηση. Ευχαριστώ πάλι για το carbon leakage και την προστασία. Μιλήσατε ξεχωριστά για την βιομηχανία παραγωγής, τη χημική βιομηχανία που είναι και βιομηχανία παραγωγής πρώτων υλών. Νομίζω κανείς εδώ εξημών δεν θα ήθελα να ανοίξει μια πόρτα ώστε η βιομηχανία αυτή να σηκωθεί να φύγει από την Ευρώπη. Θα έχουμε σύντομα και ψηφοφορία. Είχα μάλλον πρόσφατα μια ψηφοφορία εδώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και θεωρήσαμε αμφισβητήσιμη, αμφισβητήσιμο τον υπολογισμό των 30 ευρώ ανά τόνο. Είπατε ότι πράγματα πρέπει να βελτιωθούν. Πώς θα πρέπει να τροποποιηθεί η λίστα carbon leakage για να σας ικανοποιεί. Αν θέλουμε να επιτύχουμε συμφωνία για το αποθεματικό MSR, εκεί θα χρειαστούν βεβαίως πάλι συμβιβασμοί, τι θα σήμαινε για σας βελτίωση που θα, στην οποία θα μπορούσε να συμφωνήσει η χημική βιομηχανία. Να ευχαριστώ πολύ. Έχουμε και μία ερώτηση από το Ζολταν Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να μην κάνω ερώτηση αλλά μια παρατήρηση. Εκφράζω την ικανοποίησή μου για τα όσα άκουσα τον κύριο Μπότσικ γιατί για πρώτη φορά ακούσαμε κάτι από τότε που έχω γίνει ευρωβουλευτής εδώ ε, και εννοώ το εξή. Γνωρίζομαι όλοι ότι είμαστε υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος βέβαια, υπέρ της μείωσης των εκπομπών αερίων, αλλά εδώ συζητούμε πάντα μοναχά τα τεχνικά θέματα. Για την ασφάλεια της παραγωγής, για τη διαφοροποίηση κλπ. Για πρώτη φορά ήρθε κάποιος εδώ και μας, είπε, μας μίλησε καθαρά για την φτώχεια ενέργειας που πλήττει τόσους συνανθρώπους μας. Εφόσον λαμβάνουμε αποφάσεις πρέπει να έχουμε υπόψη μας και αυτό το πράγμα. Ότι και αυτό εντάσσεται μέσα στην αναζήτηση της ασφάλειας και να δούμε εάν οι καταναλωτές είναι καν εις θέση να αντέξουν τις τιμές αυτές της ενέργειας. Αν δηλαδή μπορούν να είναι, μπορεί να είναι αποδεκτό αυτό. Εμείς είμαστε στο κάτω γραφή γραφής εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών και γι' αυτό είναι σημαντικό να μην έχουμε μπροστά μας μόνο τους μακροπρόθεσμους στόχους μας αλλά και την καθημερινή ζωή των πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σιβομπέλετ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομο γιατί από ό,τι κατάλαβα θέλετε να δώσετε το λόγο και στους stakeholders σε αυτή την αίθουσα. Μια πολύ σύντομη ερώτηση στον κύριο Φόριστερ. Πώς μπορούμε να απαντήσουμε στις ανησυχίες των ενεργοβόρων βιομηχανιών Υπάρχουν ανησυχίες ότι θα υπάρχει μια έλλειψη ελεύθερης κατανομής ε, μετά από το 2021 επειδή αυξάνεται ο συντελεστής μείωσης. Ε, ξέρω ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά αυτά τα σχόλια έχουμε λάβει. Δηλαδή ακόμη και για όσους μπορούν να φτάσουν τα νέα φιλόδοξα ε, όρια, τα νέα φιλόδοξα benchmark στο μέλλον. Πώς θα αντιμετωπίσουμε κάτι τέτοιο, πώς θα απαντήσουμε σε αυτούς και πώς θα προσδώσουμε την ε, ασφάλεια, θα τους δώσουμε την ασφάλεια ότι αυτά τα δικαιώματα δεν θα είναι σε έλλειψη μετά το 2021. Ευχαριστώ. Ελπίζω να θυμάστε τις ερωτήσεις, θα ακούσουμε μία ακόμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ερώτηση μου έχει να απευθύνεται στον κύριο Μπότσεκ, γιατί εκπροσωπείται εδώ τις χημικές βιομηχανίες. Ε, υπάρχουν ε, και κάποιοι εκπρόσωποι της ΕΛ που και σας εκπροσωπείτε και θα είναι υπέρ του να ξεκινήσει το ΜΕΣΑΡ ακόμη και νωρίτερα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί η δική σας θέση είναι διαφορετική από τη δική τους, γιατί κάπως τώρα μπερδεύτηκα Δηλαδή, ποιο τμήμα της χημικής βιομηχανίας πρέπει να ακούσω. Και δεύτερον, ε, πάλι στον κύριο Μπότσο, κατευθύνεται η ερώτηση. Εδώ τώρα δεν συζητάμε την ελεύθερη κατανομή των δικαιωμάτων άνθρακα, αλλά καθώς το αναφέρατε θα ήθελα να μου πείτε επί του θέματος αυτού κάποια πράγματα, γιατί ξέρω ότι η BSF, μια μεγάλη χημική εταιρεία, μέχρι το 2013 λάμβανε ελεύθερα δικαιώματα μέχρι 5 εκατομμύρια, οπότε δεν έπρεπε να αγοράσει τίποτα. Και θέλετε να μου πείτε, όταν μιλάμε για όλα τα χημικά μέρη, πώς αυξάνεται αυτός ο αριθμός. Ευχαριστώ πολύ κυρία Άκουτ. Τώρα θα επανέλθουμε στους ομιλητές. Να προτείνω παρακαλώ στους ομιλητές μας να είναι σύντομοι για να συνεχίσουμε και τη συζήτηση. Παρακαλώ. Ο κύριος Μπότσικ, να απαντήσω πρώτα στον κύριο Γκρότε, για μένα η Carbon Leakage List δεν είναι και το θεμέλιο. Ε, εσείς ψηφίσατε κατά οποιασδήποτε παρέμβαση σε αυτήν. Μπορούμε να συζητήσουμε βέβαια για, για παράδειγμα αυτά τα benchmark πώς θα συζητηθούν μετά από την επόμενη ας περίοδο. Εκεί μπορεί να προβλεφθεί κάποια ευκαμψία ή κάποια ευελιξία. Αλλά αυτή η carbon leakage list είναι μια πολιτική ασφάλιση, α πούμε η οποία προσφέρει κάποια προστασία στους τομείς αυτούς και δεν θα πρέπει να την πειράξουμε. Μετά η ερώτηση του Bas Eichhout. Η Shell είπατε είναι υπέρ του MSR και τελείται εν συγχύσει. Και εγώ τελείω εν συγχύσει. Διότι και στον τομέα μας δεν υπάρχει και στο κομμάτι του πετρελαίου μάλλον δεν είναι όλοι σύμφωνοι. Υπάρχουν συναδελφοί μου που δεν είναι υπέρ του MSR. Πρέπει να εξετάσετε τα διαφορετικά συμφέροντα, τις διαφορετικές στρατηγικές. Οι συνάδελφοί μου της εταιρεία Shell έχουν πολλές ελπίδες από την δέσμευση και αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα. Δεν συμφωνούν άλλοι. Εγώ βέβαια, ξαναλέω, μιλώ εδώ ως εκπρόσωπος της χημικής βιομηχανίας με ευρύτατη έννοια και κατά κάποιο τρόπο και τον συνασπισμό βιομηχανιών εντάσεως ενέργειας. Η BASF είπατε δεν χρειάστηκε να, αγορήσει, να αγοράσει δικαιώματα. Είμαι βέβαιος ότι αυτό πρέπει να είναι σωστό. Αλλά τότε συγχαρητήρια στην BASF, διότι αυτό σημαίνει ότι ανταποκρίνονται στα benchmark και προφανώς έχουν πάρα πολύ ψηλή αποδοτικότητα και για το λόγο αυτό λαμβάνουν τότε δωρεάν τα δικαιώματα που ε, τους, αναλογούν. Μπράβο τους τότε. Αυτό θέλουμε άλλωστε εμείς να προσφέρουμε στις ε, βιομηχανίες που έχουν την μεγαλύτερη αποδοτικότητα τα δικαιώματα που απαιτούνται για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. We το αποτέλεσμα του MSR με βάση τις αναλύσεις που έχουμε κάνει είναι να γίνονται πιο ομαλές οι αλλαγές των τιμών. Αν ε, δεν ξαναμπούν στο σύστημα αυτή η τόνη της οπισθοβαρούς προγραμματισμού θα έχουμε περισσότερη διαφάνεια στις τιμές και αποφεύγουμε να αυξηθεί πολύ η τιμή αργότερα. Μετά από μια περίοδο δηλαδή πολύ χαμηλών ε, τιμών που σημαίνει ότι για παράδειγμα τα εργοστάσια που καίνε άνθρακα δεν έχουν περάσει σε καλύτερες τεχνολογίες. Έτσι είναι λοιπόν πιο λογική η εξέλιξη της τιμή. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, πρέπει να καταλάβουμε ότι μπορεί να έχουμε ήδη επιτύχει στην προσπάθεια μείωσης της χρήσης άνθρακα στην Ευρώπη. Και επειδή επιτυγχάνουν οι πολιτικές μας, είναι να μην έχουμε υπερβολικά λίγους τόνους. Το πρόβλημα είναι να έχουμε υπερβολικά πολλούς τόνους. Και βέβαια καμία πρόταση ενώπιών μας δεν αφαιρεί όλους αυτούς τους τόνους. Και δεν πρέπει να συγχαίουμε το MSR τόσο πολύ με τη διαρροή άνθρακα. Βεβαίως είναι πρόβλημα για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας αυτή η διαρροή άνθρακα. Αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε αυτή τη στιγμή για να τους κάνουμε παραχωρήσεις, να κάνουμε παραχωρήσεις ε, στον κλάδο, ενώ στο μέλλον έχουμε προτάσεις για να αντιμετωπιστεί το πραγματικό πρόβλημα. Πώς είναι κανείς καινοτόμος, πώς επενδύει σε καλύτερες λύσεις. Πώς δηλαδή θα συμμετέχουν όλοι στη μείωση της χρήσης άνθρακα. Όλοι προσπαθούν να προσεγγίσουν την βιομηχανία και οι περιβαλλοντολόγοι. Θα θέλαμε και εκείνοι να κάνουν μια προσπάθεια να μας προσεγγίσουν για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Άντερσον. Ο κύριος Φόρεστερ. Η ερώτηση του κυρίου Μπέλετ τώρα. Τι νομίζω για το θέμα της διαρροής άνθρακα. Πρέπει να τονίσω ότι έχουμε κοινά μέλη και με τον ε, Πίτερ. Αυτό το θέμα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι θα διορθωθεί αυτό το θέμα μέσω του MSR. Μας ενθαρρύνει ιδιαίτερα το κείμενο των ε, πορισμάτων του Συμβουλίου που λέει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα της διαρροής άνθρακα και ελπίζουμε να έχουμε ένα νομοθετικό πακέτο σύντομα που θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε και γι' αυτό. Πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε το MSR χωρίς να χάνουμε από την προοπτική μας και τα άλλα παρεμφερή προβλήματα. Και συμφωνώ με τα σχόλια του Τζέισον ότι με αυτόν τον τρόπο θα εξομαλυνθούν οι διαφορές τιμής. Θα μας βοηθήσει όλους μακροπρόθεσμα να έχουμε μια πιο σταθερή τιμή και να μην έχουμε τέτοιες ε, διακυμάνσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο, έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας. Η κυρία Σκότ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ και με τον Τζέσον και τον Τιρκ. Υπάρχει μια εξομάλυση της τιμής. Αυτό είναι το καθήκον του ΜΕΣΑΡ, του αποθεματικού και τα θέματα για τη διαρροή του άνθρακα θα πρέπει να λυθούν στο πλαίσιο της νομοθετικής δέσμας για το 2030 και το ξεκαθάρισε αυτό το Συμβούλιο. Πρέπει να είμαστε θετικοί εδώ. Λοιπόν, για τη διαρροή του άνθρακα, όπως κάποια σχόλια, αυτή η έννοια αντιμετωπίζει δύο προβλήματα. Το ένα είναι το θέμα του ενεργειακού κόστους. Ε, σε παγκόσμιο επίπεδο, ειλικρινά, δεν υπήρχε ποτέ ε, ουσιαστικά ε, ένα ίσοι κανόνες παγκοσμίω ε, και ξέρετε η γεωγραφία διαφέρει, οι Ιταλοί έχουν πολύ ήλιο, άλλοι έχουν αέριο κτλ. Ποτέ δεν υπάρχουν ίσοι κανόνες παγκοσμίω, η Ευρώπη δεν είναι και σε πολύ καλή κατάσταση εδώ. Πρέπει λοιπόν να ακολουθήσει μια διαφορετική στρατηγική από τις τακτικές αυτών που έχουν πολύ φτηνή ενέργεια. Και εδώ εντάσσεται η ενεργειακή αποδοτικότητα. Ένα άλλο θέμα είναι ο ανταγωνισμός για τις επενδύσεις. Και εδώ υπάρχει και ένα θέμα και για το δικό μου κλάδο. Τώρα είμαστε πολυεθνικές εταιρείες, πολλοί από εμά και επενδύουμε εκτός της Ευρώπης. Και αυτό το μοντέλο βλέπω ε, στον σε μεγάλες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας τώρα έχουν περισσότερους ε, πελάτες ε, στη Τουρκία παρά στη Γερμανία και έχουν περισσότερα περιουσιακά στοιχεία στη Ρωσία, στη Βραζιλία. Επενδύουμε εκτός της Ευρώπης γιατί δεν ξέρουμε τι να κάνουμε εντός της Ευρώπης γιατί δεν υπάρχει πολιτικό μήνυμα και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε. Αυτό είναι το λογικό. Νομίζω και οι συνάδελφοι από τη ΣΕΛ ε, θα με συγχωρήσουν να πω ότι είναι μια πολύ ευφυής εταιρεία και σίγουρα θα έχει ηγετικό ρόλο σε 100 χρόνια. Εγώ θα έπαιρνα πάρα πολύ σοβαρά οποιαδήποτε θέση αναπτύξουν για οποιαδήποτε πολιτική. Μάλιστα, εδώ είμαστε. Υπάρχει και επικύρωση, λέει ο πρόεδρο. Έχουμε ακόμα 10 λεπτά. Ο κ. Μιλσταρτέλης θέλει να κάνει μια ερώτηση. Ευχαριστώ. Με την διαρροή του άνθρακα και πάλι, πιθανότατα έχει να κάνει. Έχουμε μία μελέτη από για να κάνουμε μία σύγκριση σε σχέση με το MSR και τι άλλο θα μπορούσε να υπάρχει. Έχετε κάποια σχετική πληροφορία. Ή ε, θα μπορούσατε να μας πείτε ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των δύο προσεγγίσεων. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα δώσουμε το λόγο στο πίσω μέρος της ε, αίθουσας. 30 ε, δευτερόλεπτα, αν είστε πολύ καλοί, θα έχετε κι άλλοι το λόγο. Και πιθανότητα θα δώσουμε ένα λεπτό στους ε, ομιλητές μας για να απαντήσουν. Και αν θέλετε μπορείτε να στείλετε την ερώτησή σας και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ο κύριος Μόρισον, 30 δευτερόλεπτα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ερώτησή μου είναι για τον κύριο Μπόρτσεκ εγώ εκπλήσωμαι που δείχνει κάποια, κάποιο δισταγμό για να δεκτεί μια έγκαιρη νωρίτερη εφαρμογή του MSR, καθώς ε, ο τομέα των χημικών βιομηχανιών έλαβε 28 εκατομμύρια δικαιώματα το 2013 και εμείς υπολογίσαμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε αύξηση 20% στις εκπομπές χωρίς να χρειαστεί να αγοράσει κανείς ούτε ένα δικαίωμα. Έτσι λοιπόν, γιατί ο χημικός τομέας μυθεί τα ελεύθερα δικαιώματα, τα δωρεάν δικαιώματα που δεν χρειάζεται. Μόνο 11 δευτερόλεπτα παραπάνω από το χρόνο σας. Παρακαλώ, εκεί στο πίσω μέρος της αίθουσας. Ε, συγγνώμη, πρέπει να με βοηθήσετε να μου πείτε το όνομά σας. Σας ευχαριστώ. Η ερώτησή μου είναι για τον κύριο Τάνκαν. Ε, πιστεύετε ότι αν έχουμε μία ταχεία έκβαση του MSR θα μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα άπαξ και διαπαντός ότι αφορά την διαρροή του άνθρακα μέσω του πακέτου για το 2030. Μάλιστα, πολύ εντυπωσιακή ερώτησή σας, πολύ γρήγορη. Κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Αν όχι, να περάσουμε στα μέλη του πάνελ. Να ξαναρχίσουμε τώρα από τα δεξιά προς τα αριστερά. Κυρία Σκότ, αν μπορείτε ξεκινήστε. Νομίζω ότι θα συμφωνούσα μαζί συντομότερα λειτουργήσει το MSR, θα προτιμούσαμε του χρόνου, τόσο πιο θα προχωρήσει και η δέσμη μέτρων για το 2030. Δεν νομίζω ότι θα η διαδικασία της συναπόφασης θα κρατήσει μόνο 11 μήνες. Νομίζω ότι μάλλον θα κρατήσει δύο χρόνια και παραπάνω και αν δούμε τα αριθμητικά στοιχεία φτάνουμε πολύ κοντά στο 2020. Το συντομότερο το καλύτερο λοιπόν. Τώρα για τον τομέα του Χάλιβα. Πραγματικά το συμπονώ, γιατί είναι ένα τομέα που αντιμετωπίζει τέτοιε προκλήσει όπω και εμεί ε, στον τομέα τη ηλεκτρική ενέργεια. Αλλάζει η αγορά, αλλάζουν τα επιχειρηματικά μοντέλα και μπορώ να πω ότι η αντίδραση που είχαμε είναι να αποφασίσουμε ότι πρέπει να πάμε μπροστά από αυτέ τι αλλαγέ και να επενδύσουμε στην κοινοτομία. Πολύ ωραία. Παρακαλώ, κύριο Φόριστερ. Εδώ θα ακούσετε μια χοροδία υποστήριξης, μια ομοφωνή υποστήριξη για ταχεία δράση. Γιατί μπορεί να φαίνεται ότι ε, το MSR να έρχεται ταχύτατα, αλλά εμείς αυτές τις πληροφορίες τις έχουμε εδώ και πολύ καιρό, έχουμε αναλύσει όλο αυτό το θέμα λεπτομερώς και νομίζω ότι από τη δική μας σκοπιά είναι καιρός να αναλάβουμε δράσεις. Αλλά βέβαια πρέπει να διατηρήσουμε μία εστίαση στο επόμενο μεγάλο ζήτημα που θα είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, ίσως και πιο σημαντικό. Και αφορά τα στοιχεία της νομοθετικής δέσμης του 2030. Μάλιστα. Εσείς ο, οι οδηγίε που έδωσε ο κ. Ιούνκερ για στον Αρία Κανιέτε είναι να προωθήσει την ε, νομοθεσία σύντομα στην αρχή της θητείας του και ελπίζουμε να συμβεί αυτό και να μην ανακόψει την πορεία αυτή το MSR που είναι μεν σημαντικό αλλά είναι απλώς ένα ε, βήμα αναγκαιωμένο όχι επαρκές. Υπάρχουν και όλα τα άλλα μέτρα του πακέτου 2030 και θα βλάψει πολύ την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών θεσμών μέσα στην Ευρώπη και αυτούς που επιδιώκουν την υιοθέτηση των ανανεώσιμων ε, ενεργειών κτλ. Εάν αυτό το συγκεκριμένο αντικείμενο συναπόφασης ανακόψει την πορεία όλης της υπόλοιπης νομοθεσίας που είναι αναγκαία. Και τέλος ο κ. Μπότσεκ. Σας ευχαριστώ. Το σύστημα ETS υποτίθεται ότι θα συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου μείωση των ε, εκπομπών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Με το MSR τώρα αλλάζουμε το σύστημα και πάμε να πετύχουμε το στόχο με ένα συμφωνημένο κόστος. Πρόκειται για συστημική αλλαγή. Αναρωτηθείτε αν πραγματικά αυτό θέλετε. Για να απαντήσω στην ερώτηση του Ντάμιαν, οι βιομηχανίες έντασης ενέργειας δεν εμπορεύονται εκπομπές. Δεν είναι αυτή η δουλειά τους. Η δουλειά μας είναι να φτιάχνουμε προϊόντα, να παράγουμε προϊόντα για τους πελάτες μας. Και το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, κάποιες φορές και κάποιοι τομείς, έχουν υψηλές κατανομές δικαιωμάτων. Είναι αυτό είναι λυπηρό, δεν είναι αυτό που επιζητήσαμε εμείς από την αρχή. Θα το θυμάστε, από την αρχή είχαμε ζητήσει εμείς εύκαμπτη κατανομή, διότι το βλέπαμε να έρχεται το πρόβλημα. Ότι ή θα υπάρξει κρίση και επομένως υπερπροσφορά ή σε περίπτωση ανάπτυξης θα υπάρξει μειωμένη προσφορά, δηλαδή ελληματική προσφορά και επομένως θα αυξηθούν οι τιμές. Εκεί πρέπει να παίξει το ρόλο της ευκαμψίας. Βεβαίως πάντοτε υπό τον όρο ότι αυτοί που αποδίδουν περισσότερο έχουν επαρκή δικαιώματα για να κάνουν τη δουλειά τους και ότι υπάρχουν πάντοτε και επαρκή δικαιώματα για δωρεάν κατανομή. Και αν φτάσουμε σε ένα μοντέλο όπου αυτός ο μηχανισμός σταθερότητας της αγοράς που μπορεί να έχει και άλλο όνομα αν μπορέσουμε να το μετατρέψουμε το μηχανισμό αυτό σε ένα εργαλείο που θα επιτρέψει την δωρεάν κατανομή, τότε βρισκόμαστε σωστή πορεία. Ευχαριστώ κύριε Μπότσοκ. Με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω ολόκληρο το πόνελ Μπότσοκ και τους υπόλοιπους κυρίους και την κυρία. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχιστεί η συζήτηση. Τώρα θα δώσω με μεγάλη χαρά τον λόγο πάλι στον Ιβο Μπέλετ ο οποίος θα συνεχίσει την ίδια συζητήσεως για το, υπόλοιπο, για το τελευταίο τμήμα της. Αν θέλει λοιπόν το πάνελ παρακαλώ να κατέβει στα έδρανα. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους εμπειρογνώμονες. Καταληκτικές παρατηρήσεις. Τελικό δεκάλεπτο. Χαιρετίζω τον Ζος Ντελμπέκε. Μας υποσχέθηκε ότι θα έρθει και ήρθε πρώτα απ' όλα. Ήταν η πρώτη επίσημη συνάντηση της Νέας Επιτροπής. Πήγε καλά κύριε Ντελμπέκε. Ωραία. Ο κύριος Ντελμπέκε όπως ξέρετε, είναι Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης για την Κλιματική Δράση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα παρουσιάσει την άποψη της Ευρωπαϊκής και έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιβο Μπέλετ. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ και ευχαριστώ θερμά που οργανώσατε αυτό το σεμινάριο. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε βαθύτερα περί τίνος πρόκειται. Και επειδή ήμουν παρόν σε ένα τμήμα της συζήτησης, νομίζω ότι επιτύχατε σε αυτή την προσπάθεια. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσει το ETS να παίξει σωστά το ρόλο του. Ακούσατε τι είπαν οι αρχοί κρατών κυβερνήσεων πριν από 10 μέρε. Είναι σαφής στήριξη του ETS. Είναι το συστατικό κλειδί για να μειώσουμε τα αέρια θερμοκηπίου. Στην προπτική του 2030 υπόθηκε επίσης ότι πρέπει να μεταρρυθμιστεί το ETS της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να σταθεροποιηθεί η αγορά όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σαφής λοιπόν η σημασία της συζήτησης σήμερα και με ενθαρρύνουν ιδιαίτερα αυτά που θα μπορέσω να συνοψίσω και να μεταφέρω στις υπηρεσίες μου. Τα εξής πέντε. Πρώτον, βοηθάει πολύ αυτή η συζήτηση, αλλά βλέπω ότι υπάρχει και πολλή στήριξη για την ε, γενική προσέγγιση της Επιτροπής. Δηλαδή ένα σύστημα που να βασίζεται σε κανόνες, όχι με διακριτική ευχαίρεια συμμετοχή ή όχι. Ένα σύστημα που να βασίζεται στην προσφορά, που να μην παρεμβαίνει άμεσα στις τιμές. Ένα σύστημα προσφοράς πρέπει να το χειριστούμε με κάποιες παραμέτρους. Ορισμένοι θέλουν πιο φιλόδοξες τιμές για αυτές, άλλοι πιο προσεκτικές. Νομίζω όμως ότι η πρόταση της Κομισιόν ε, είναι ακριβώς ε, μια μετριοπαθή στη μέση μεταξύ των ακραίων αυτών προσεγγίσεων με βάση και τις ε, εξομοιώσεις που κάναμε και που θα βρείτε στο site μας. Δεύτερον, αυτό που ήδη υπόθηκε, ότι το χρονοδιάγραμμα για να ολοκληρώσετε κι εσείς ως συνομοθέτες την εργασία αυτή είναι πολύ σημαντικό. Γιατί δεν έχει έννοια να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε ένα μέσο που δεν τα πάει καλά. Πρέπει λοιπόν να είναι αποδοτικός, λειτουργικός αυτός ο μηχανισμός γιατί αυτό θα αυξήσει την εμπιστοσύνη των ε, συμμετεχόντων στην αγορά, θα αυξήσει τη σταθερότητα της αγοράς άνθρακα, θα είναι το σωστό μήνυμα που δίνουμε στους επενδυτές και ξέρετε ότι ο νέος πρόεδρος, κ. Γιούνκερ, ανήγγειλε εδώ ότι θέλει ένα πακέτο επενδύσεων 300 δις, το οποίο θα υποβληθεί σύντομα. Και τμήμα αυτών των επενδύσεων θα είναι σε τομείς που είναι πολύ σημαντικοί για τα θέματα που συζητάμε. Για τον ενεργειακό κλάδο θέλουμε να κάνουμε επενδύσεις εκεί και τον τομέα των μεταφορών. Πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε αυτό το πακέτο των 300 δις. Όσο ταχύτερα λοιπόν εισαχθεί, ολοκληρωθεί μάλλον, αυτή η πρόταση για το MSR, τόσο καλύτερα. Εμείς έχουμε κάνει το δικό μας τμήμα της δουλειάς μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου, αλλά φυσικά πρέπει να καταλήξουμε σε αυτό το μηχανισμό. Αυτό θα μας βοηθήσει στην περαιτέρω εργασία μας και στις περαιτέρω προτάσεις που θέλουμε να υποβάλουμε. Σημαντικό λοιπόν το χρονοδιάγραμμα. Και νομίζω ότι η συζήτηση που μόλις έλαβε χώρα θα επιτρέψει στους συνομοθέτες να περάσουν στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων. Τρίτον, ένα σχόλιο για τη διαρροή άνθρακα. Ακούσαμε τα υπέρ και τα κατά. Θέλω να υπογραμμίσω γορηματικότατα, αυτό που είπαν και αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων. Υπάρχει μία πλήρης και μακροσκελής παράγραφος, αλλά στέλνει και το βασικό μήνυμα το κείμενο, ότι θα υπήρχε πολύ μεγαλύτερη ανησυχία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων σε αυτό το τομέα αν δεν είχε υπάρξει αυτή η παράγραφος. Γιατί όλα τα μέτρα που υπάρχουν θα ε, πάψουν σταδιακά να ισχύουν μέχρι το 2027 και αυτές οι διαβεβαιώσεις που δόθηκαν από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων είναι ότι το σύστημα των ελεύθερων χορηγήσεων θα διατηρηθεί, θα βελτιωθεί, θα πρέπει να γίνει πιο αποδοτικό, αλλά στα βασικά του στοιχεία το σύστημα αυτό θα συνεχίσει να εφίσταται. Και αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής του συστήματος και θα το λάβει υπόψη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις προτάσεις που θα υποβάλει για το ETS μετά την έγκριση του πακέτου για το 2030. Τέταρτον, αλληλεπίδραση μεταξύ ETS και άλλων ε, μηχανισμών πολιτικής, για παράδειγμα για τις ανανεώσιμες και την αποδοτικότητα της ενέργειας. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις για το εάν και κατά πόσον ένα από τα μέσα μας πρέπει να κυριαρχεί. Νομίζω ότι με την έγκριση του MSR η συζήτηση αυτή θα λήξει μια για πάντα. Και το χαιρετίζω πολύ αυτό. Γιατί πολλές φορές ε, υπήρχαν διαφορετικές ερμηνείες για το ποια είναι η ε, πρόθεση του Α ή του Β τμήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο μηχανισμός αυτός θα μας επιτρέψει να, να επιτύχουμε συνεργασία και κοινή δράση των διαφόρων πλευρών του συστήματος. Το MSR θα αφορά την ε, ζήτηση. Οποιασδήποτε λοιπόν ε, επιπλέον δυνατότητες θα προκύψουν λόγω βελτίωσης αποδοτικότητας για παράδειγμα θα αντιμετωπιστούν από το μηχανισμό αυτό. Αυτό θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε εκρεμή προβλήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή και θα είναι μια ανακούφιση για όλους μας. Ορισμένα σχόλια που ακούμε τώρα θα πάψουμε να τα ακούμε οριστικά. Και τέλος, η συζήτηση για ε, νωρίτερη εισαγωγή. Η Επιτροπή προτείνει 2021. Για μια σειρά από λόγους, καλούς κακούς. Θα θυμάστε ότι όταν ε, εκπονήσαμε την πρότασή μας, ε, η συζήτηση για τον όπιστο βαρύ προγραμματισμό ήταν πολύ έντονη. Δεν θέλω να επανέλθω, αλλά είπαμε σαφώς ότι εάν οι συνομοθέτες θέλουν νωρίτερη εισαγωγή, συμφωνούμε. Και Εάν ε, οι οπισθοβαρείς χορηγήσεις πάνε κατευθείαν στο αποθηματικό, αυτό θα ε, καθησυχάσει τους πάντες ότι θα υπάρχει περισσότερη σταθερότητα τιμών και όχι διακυμάνσεις. Θετικά λοιπόν θα αντιμετωπίζαμε την νωρίτερη εισαγωγή και όποιος διαβάσει την μελέτη αντικτύπου μας θα δει ότι Μία από τις αναλλακτικές λύσεις που εξετάσαμε ήταν ακριβώς η νωρίτερη εισαγωγή. Καταλήγω λοιπόν, τονίζοντας ότι ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η συζήτηση, αναφέρθηκαν όλα τα βασικά θέματα που αφορούν τη συζήτηση αυτή και ελπίζουμε ιδιαίτερος στο Συμβούλιο ξέρουμε ότι έχει αρκετά προχωρήσει η δουλειά αλλά πιστεύουμε ότι και οι επικείμενες συνεδριάσεις ΕΝΒΙ και ΙΤΡΕ θα πάνε σε βάθος, θα βοηθήσουν. Ίσως λοιπόν θα μπορούσαμε ήδη να σκεφτούμε τι συμβιβασμούς θα μπορούσαμε να επιδιώξουμε για να διευκολύνουμε τους τριμερείς διαλόγους που θα χρειαστούμε αργότερα. Όσο καλύτερα προετοιμάσουμε την εργασία μας και τη δική σας εδώ στις επιτροπές σας, τόσο ταχύτερα θα καταλήξουμε και από πλευρά του νέου μου επιτρόπου, τον οποίο θα συναντήσετε προσεχώς, από πλευράς λοιπόν και του νέου επιτρόπου μας, καλωσορίζουμε ιδιαίτερος αυτές τις συζητήσεις και προσβλέπουμε σε μια ταχεία κατάληξη των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ πολύ. Και εύχομαι κάθε επιτυχία στην επόμενη φάση της εργασίας σας για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ, Σασταλμπέκης, και φαντάζομαι θα συναντηθούμε και πάλι στο εγγύ μέλλον. Τελικέ παρατηρήσεις ε, για δύο λεπτά. Αγαπητοί φίλοι, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι το σύστημα εμπορία εκπομπών χρειάζεται μια διαρθρωτική μεταρρύθμιση, μεγαλύτερη συνέχιση, να λειτουργεί λιγότερο, αστα... με λιγότερο σταθή τρόπο η αγορά. Όλα αυτά τα αιτήματα διατυπώθηκαν σε αυτό το εργαστήριο. Φυσικά υπάρχουν πολλά εκκρεμή ζητήματα, αναφέρθηκε ο κύριο Στεμπέλ και φυσικά το χρονοδιάγραμμα είναι σημαντικό. Μιλήσαμε για το 2021 ή για μια πιο έγκαιρη έναρξη και φυσικά τα αποστοβαρή δικαιώματα σχετίζονται και με το χρονοδιάγραμμα, η συνέχιση και η βελτίωση των διατάξεων ε, για τη διαρροή του άνθρακα είναι εκτός ε, του άμεσου πεδίου εφαρμογή αυτής της ε, απόφασης, αλλά φυσικά υπάρχει στενή σύνδεση. Και άλλη μια πτυχή είναι το θέμα των κατοφλίων και των παραμέτρων του MSR. Δεν υπάρχει ακόμα ευρεία συνένεση. Παρ' όλα αυτά θα συνεχίσουμε έντονες διαβουλεύσεις με τους περισσότερους από εσά τις επόμενες εβδομάδες. Και Είμαστε αισιόδοξοι και ελπίζουμε ότι θα καταλήξουμε σε έναν ισορροπημένο συμβιβασμό. Ίσως ε, και κάτι ακόμη για το χρονοδιάγραμμα στο Κοινοβούλιο. Από εδώ και πέρα ο κύριος Τελμπέκε θα επιταχύνει τις δραστηριότητες εδώ στο Κοινοβούλιο. Πρώτη ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή ΕΝΒΗ έχει προγραμματιστεί για τις 3 Δεκεμβρίου. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι ταχύτητα της 11 Δεκεμβρίου και οι συνάδελφοι στην Επιτροπή Ήτρε θα συζητήσουν στις 17 Νοεμβρίου και θα ψηφίσουν στις 21 Ιανουαρίου. Και εδώ η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας έχει σχεδιαστεί για τις 23 ή 24 Φεβρουαρίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολλού ανθρώπου. Καταρχήν του φίλου μα από την Ιταλική μόνιμη αντιπροσωπεία, με του οποίου συνεργαστήκαμε πολύ στενά τι τελευταίε εβδομάδε και θα συνεχίσουμε φυσικά και τι επόμενε εβδομάδε, γιατί υπό την Ιταλική Προεδρία το Συμβούλιο έχει σημειώσει πολύ μεγάλη πρόοδο. Σα ευχαριστούμε λοιπόν. Γι' αυτό και συγχαρητήρια. Η Λετωνία θα αναλάβει την Προεδρία από τον Ιανουάριο και ελπίζω ότι θα μπορέσει να ολοκληρωθεί μεταρρύθμιση υπό την Λετωνική Προεδρία. Θέλω να ευχαριστήσω ένθερμα όλους τους ομιλητές, όλα τα μέλη του πάνελ. Ευχαριστώ πολύ τον Ματίας Γκρότη, τον Ιαν Ντάνκαν που ήθελα να συμπροεδρεύσουν σε αυτό το εργαστήριο. Ευχαριστώ και το ε, Τμήμα Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ και την Γραμματεία που μας βοήθησε εδώ στη διοργάνωση και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς. Ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να σας ξαναδώ σύντομα. Καλό σας βράδυ.